ζητήσω από τον τύπο να ολοκληρώσει τις εργασίες του για να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ καθίστε λοιπόν. Να ησυχάσει η αίθουσα. Θα τεθούν πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα. Θα ακούσουμε και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν με τις κάμερες να φύγετε για να ξεκινήσουμε. Can I ask everyone at the back, please? Επίσης, να ζητήσω να καθίσετε όλες τις θέσεις σας και εσείς εκεί πίσω. Και λίγη ησυχία. Okay. Thank you very much indeed. Uh, so, ladies and... Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. για να ξεκινήσουμε τη σημαντική αυτή ακρόαση. Είναι λοιπόν ε, μεγάλη μου χαρά ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Καταναλωτή και της ε, να καλωσορίσω τον Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι υποψήφιος επιτροπός για την ιστορική αγορά, την ακρόαση του οποίου θα, θα ακούσουμε σήμερα το απόγευμα. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τις οδηγίες για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψήφιους βάσει των δεξιοτήτων του και της γενική τους ε, ικανότητας και αξιολογεί και την ικανότητά τους για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αυτός είναι ο στόχος των, της τρίτης ακρόασης σήμερα το απόγευμα. Και ίσως θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε την σημερινή ακρόαση αναφέροντας το, την επιστολή αποστολής που έστειλε ο κύριος Μπαρόσο προς τον κύριο Μπαρνιέ για την ανακοίνωση της υποψηφιά του και αναφέρει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει ε, πολιτική κατεύθυνση και να προάγει το έργο της. Και στο πλαίσιο αυτό ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα είναι υπεύθυνο για να δώσει μια νέα όθηση στην ενιαία αγορά, προωθώντας τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες, τις δημόσιες προμήθειες, την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και των επαγγελματικών προσόντων. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πολλά σχετικά σχόλια σήμερα το απόγευμα. Η δομή της ακρόασης θα είναι η εξής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είναι σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου η συνάδελφος Άρν που είναι ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου θα αναλάβει την Προεδρία. Έτσι λοιπόν θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ε, ακρόασης. Θα καλέσουμε τον κύριο Μπαρνιέ να κάνει μια εισαγωγική δήλωση. Μετά θα έχουμε μία ώρα και 20 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες της Επιτροπής Ιστορικών Υποθέσεων, Ιστορικής Αγοράς. Και για κάθε ερώτηση θα έχουμε ένα λεπτό. Ο Επίτροπος θα απαντήσει δύο λεπτά και ύστερα θα έχουμε ένα λεπτό πάλι ερώτηση και ένα λεπτό απάντηση. Θα είμαι πολύ αυστηρός και εγώ και η κυρία Μπόιλς σε ό,τι αφορά το χρόνο ομιλίας. Ήμασταν άλλωστε και χτες για να προχωρήσουμε γρήγορα και να καλέσω τους ε, συναδέλφους μου να θέτουν συγκεκριμένα και γρήγορα ερωτήματα. Το ίδιο ισχύει και για τις επιρωτήσεις και στο τέλος θα κάνει κάποια τελικά σχόλια ο Επίτροπος προτού περάσουμε στο επόμενο τμήμα της ε, συνάντησης. Να σας επενθυμίσω επίσης ότι ε, η ακρόαση αυτή μεταδίδεται και στο διαδίκτυο και θα μεταδοθεί και στην ε, τηλεόραση αργότερα. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Είναι μεγάλη μου λοιπόν τιμή και χαρά και προσκαλώ τον υποψήφιο επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, που βρίσκεται στη μεταβατική φάση. Αν θέλετε, από τα έντρανα της Επιτροπής στα έντρανα εδώ μπροστά γιατί ήταν μέλος τους τελευταίους έξι μήνες της Επιτροπής μας. Τώρα λοιπόν μας βλέπετε από την άλλη πλευρά. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν βρίσκομαι στην ίδια θέση, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι στην ίδια αίθουσα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι μπροστά σας σήμερα ως πολιτικός άνδρας, ο οποίος απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες πολιτικούς. Πολιτικός άνδρας που γνωρίζει τη σημασία της δημοκρατικής νομιμότητας, τη σημασία της εργασίας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ο οποίος εδώ και καιρό, όπως και εσείς, έχει ευρωπαϊκή δέσμευση και θα είμαι πάντα υπόλογος. Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την ακρόαση που είναι μια απαιτητική στιγμή με κάπως πιο προσωπικά σχόλια. Με σημάδεψε το όχι του γαλλικού δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το 2005. Με εντυπωσίασε πολύ με σημάδεψη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την αποτυχία. Αλλά κυρίως για μένα αυτή η αποτυχία ήταν η έκφραση μιας δυσαρέσκειας που συμμερίζονται πολλοί λαοί πέραν της Γαλλίας. Ήταν η απόδειξη ότι η Ευρώπη απομακρύνθηκε από τους πολίτες. Το ευρωπαϊκό όμως σχέδιο αυτό των πατέρων της Ευρώπης είχε ακριβώς στην καρδιά του την οικοδόμηση της μεγάλης κοινή αγοράς, της κοινή οικονομικής μας και κοινωνικής ζωής. Πώς να το πω αλλιώς. Είναι αυτή η βούληση να είμαστε μαζί που τροφοδοτείται από το συμφέρον του να είμαστε μαζί. Με την δυνατότητα δράσεως που θα κρίνατε να μου δώσετε και με την εμπιστοσύνη του Προέδρου Μπαρόζο, η φιλοδοξία μου και η στρατηγική μου για αυτά τα πέντε χρόνια θα είναι να συμφιλιώσω ξανά αυτήν την βούληση να είμαστε μαζί και την αναγκαιότητα να είμαστε μαζί σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν στην καρδιά της ενιαίας αγοράς πρέπει να βάλουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, αυτούς που το ζουν καθημερινά. Σε αυτό το πρώτο τμήμα, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στις αδυναμίες. Ο Μάριο Μόντι, που ακούσατε πριν από μερικές εβδομάδες στην Επιτροπή ΙΝΚΟ, αναφέρθηκε στην κούραση της εσωτερικής αγοράς. Η φιλοδοξία μου, κυρίες και κύριοι, είναι να σας προτείνω να δώσουμε μια νέα όθηση για τα επόμενα πέντε χρόνια στην εσωτερική αγορά έναντι της κρίσης ξαναείδαμε το συμφέρον του να είμαστε μαζί και όχι ο καθένας μόνος του. Προσοχή όμως. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση αυτή τη στιγμή ενισχύει τις πιέσεις ώστε όλες οι κυβερνήσεις να δώσουν εθνικές απαντήσεις, βραχυπρόθεσμες, μερικές φορές απαντήσεις κλεισίματος. Όμως γνωρίζουμε ότι ο κατακαιρματισμός του της αγοράς είναι φρένο στην ανταγωνιστικότητα και σε πολλούς τομείς έχουμε κοινού κανόνες, όμως δύσκολα τους εφαρμόζουμε κατά κοινό τρόπο. Όλα αυτά δημιουργούν εμπόδια στις ανταλλαγές, εμπόδια για τις επιχειρήσεις και έλλειψη κατανόησης από τους πολίτες. Σας προτείνω μαζί να προσπαθήσουμε ώστε να μειώσουμε αυτά τα εμπόδια. Να παγιώσουμε σας προτείνω και να επιτύχουμε μαζί την μετάβαση που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια με την όθεση του Ζακ Ντελόρ από το εθνικό καθένας και απάνω του στο ευρωπαϊκό όλοι μαζί. Προτείνω αυτή την εσωτερική αγορά να την θέσουμε στην υπηρεσία της νέας στρατηγικής για το έτος 2020 του Μανουέλ Μαρόζο Γι' αυτό μαζί σας θέλω να αναπτύξω και ακούγοντας όλους την δράση μου ανάμεσα σε πέντε προτεραιότητες την εμπιστοσύνη που πρέπει να ενισχύσουμε στην προστασία που δίνει η εσωτερική αγορά. Δεν είναι γραφειοκρατική εφεύραση η ενιαία αγορά. Είναι η δική μας αγορά και αφορά την καθημερινή ζωή. Πρέπει να δώσει υπηρεσίες και αγαθά ασφαλή, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Να επιτρέψει στις επιχειρήσεις και στους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Το δικαίωμα της κατανάλωσης, ελεύθερα και με εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίντερνετ πολλαπλασιάζει τις προσφορές και θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την ανάπτυξη θεσπίζοντας ένα ασφαλές πλαίσιο που δίνει τις απαραίτητες εγγυήσεις στον καταναλωτή. Το δικαίωμα να εργαστεί κανένας και να ζει σε άλλη χώρα πέραν της δικής του και να αναγνωριστούν τα προσόντα του. Τα κράτη-μέλη έπρεπε εδώ και δύο χρόνια να ενσωματώσουν την οδηγία του 2005. Πολλοί δεν το έκαναν ακόμα και αυτό είναι εις βάρος της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. 20% των προβλημάτων που υποβάλλονται στο δίκτυο Solvit ακριβώς αφορούν αυτό το θέμα. Θα αναλάβω εκεί τις ευθύνες μου. Και αν πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, να συνεργαστούμε δηλαδή με τους απαραίτητους τομείς για να δώσουμε στους Ευρωπαίους την επαγγελματική κάρτα που επιμένουν. Δικαίωμα λοιπόν για τις επιχειρήσεις και κυρίως και πρώτα για τις ΜΜΕ να, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να α, εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες. Θέλω να περάσουν όλα τα νομοθετικά κείμενα για την ενιαία θηρίδα και την, γραφειο... την ε, διοικητική συνεργασία. Μια δεύτερη προτεραιότητα θα είναι να αξιοποιήσω την ε, δημιουργία και την καινοτομία. Πλούτος μας είναι οι άντρες και οι γυναίκες, ο πολιτισμός τους στην Ευρώπη, στον πληθυντικό, η καινοτομία τους και η δημιουργικότητά τους. Δεν θα διστάσουμε να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους δημιουργούς για τα έργα τους. στον ψηφιακό κόσμο που βρισκόμαστε όμως, η γνώση και το περιεχόμενο γίνονται προσβάσιμα σε μεγάλο αριθμό. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε το πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων και από κοινού καλύτερα να διαχειριστούμε τα δικαιώματα στο ίντερνετ και για τα ορφανά έργα. Αν έχουμε τέτοιου είδους ελκυστικό περιεχόμενο θα μειώσουμε την πειρατεία. Το ίδιο θα κάνουμε για την προστασία των βιομηχανικών καινοτομιών. Το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουμε κοστίζει ακριβά και θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα και να κινητοποιήσουμε τις απαραίτητες τεχνολογίες. Και μπορούμε να εξετάσουμε ένα κανονισμό για το θέμα το γλωσσικό και να προτέσουμε και το θέμα της δικαιοδοσίας. Μιλάμε για καινοτομία και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά είναι, αμφισβητούνται από τις ε, απομιμήσεις που είναι εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θέλουμε να αναπτύξουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά των Απομιμήσεων και θέλουμε να έχουμε ένα ε, μεγαλύτερο φάσμα κυρώσεων και στην Ευρώπη αλλά και στους κυρίους εταίρους μας και αυτό θα το κάνουμε με τον συνάδελφο που είναι επιφορτισμένος για την καταπολέμηση της απάτης. Τρίτη προτεραιότητα θα είναι οι πολίτες να είναι στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς. Είναι πρόκληση για όλους τους επιτρόπους να δώσουν έννοια στο ευρωπαϊκό μοντέλο της ε, κοινωνίας. Για μας εδώ αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της αγοράς θα πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη πρόοδο και όχι το ανάποδο. Βελτιώνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικέ υπηρεσίες να μπορούν οι πολίτες να αναπτέξουν τις γνώσεις τους και το πολιτισμό του. Θα εξετάσω τη δυνατότητα να έχουν τα ιδρύματα και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ένα ευρωπαϊκό καθεστώς. Θα εξετάσουμε το μοντέλο των, ε, ε, των οργανώσεων αλληλοβοηθείας Θέλουμε λοιπόν ένα, ε, μια, ένα νόμο που να μπορέσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να είναι κερδοφόρες και ταυτόχρονα καταπολεμούν τον αποκλεισμό. Και τέταρτη προτεραιότητα, η εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι παρούσα σε αυτήν τη νέα ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Πιο οικολογική, βιώσιμη και θα χρησιμοποιήσω το εύνομο όπως και το άρθρο 9 της Συνθήκη της Λισαβόνας για τις μελέτες κοινωνικής επικτότητας και περιβαλλοντικής, ε, ε, περιβαλλοντικών διαδικτύπου για να εξετάσουμε τις οδηγίες. Και θα πρέπει καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο δις, το 2-3 των ε, κρατικών προμηθειών για να ενθαρρύνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Επίσης αναφέρομαι και στη σύστασή σας για την ε, αμοιβή των διοικητών. Δεν αφορά μόνο τις τράπεζες αλλά και τις ε, βιομηχανίες. Τέλος, πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους επιτροπούς για να δούμε τις σχέσεις διανομής, τη σχέση ανάμεσα σε παραγωγό και τη διανομή, την πρόσβαση στο εμπόριο και το δίκαιο εμπόριο. Κυρίες και κύριοι, αυτές οι, αυτοί είναι οι προσανατολισμοί με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ μαζί σας, με το Συμβούλιο Υπουργών σε διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΙ και είμαι τώρα έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Well, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Σα έδωσα λίγο χρόνο παραπάνω και προειδοποιώ του υπόλοιπου ομιλητέ ότι δεν πρέπει να το κάνω και για αυτού Να περάσουμε στι ερωτήσει και να δώσω το λόγο στον Ανδρέα Φάπτο τον Ιστή από το ΕΛΚ και την Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς, το λόγο. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ υποψήφιοι επίτροπε, σας εκτίμησα ιδιαίτερος ως μέλος αυτής της Επιτροπής του Κοινοβουλίου και με χαρά σας είδα να φτάνετε στην Επιτροπή στο χαρτοφυλάκιο το πιο σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή μας περιγράψατε με εντυπωσιακό τρόπο τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια μαζί μας στην Ευρώπη. Αλλά κατά το παρελθόν είχα κάποιες ε, συζητήσεις και έχω διαβάσει και κάποια κομμάτια σας για τις πολιτικές σας ε, προτεραιότητες. Και όλοι μας έχουμε το πολιτικό μας παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς ε, θα κλιμακώσετε αυτές τις προτεραιότητές σας και θα ήθελα να σιγουρευτώ ότι δεν θα επηρεαστείτε από κανένα πολιτικό κόμμα τα επόμενα χρόνια, αλλά ότι θα θέσετε όλες τις ε, προσπάθειες για να εξυπηρετήσετε τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. θα ξεχάσω την ποιότητα των εργασιών που κάναμε από κοινού σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Τώρα που την εγκαταλείπω για να γίνω επίτροπος χάρη στην έγκρισή σας αν αυτή γίνει, δεν θα την ξεχάσω. Ούτε θα ξεχάσω και την σωστή προεδρία σας της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σουάμπε, αναφέρθηκε στην πολιτική μου δέσμευση. Εγώ είμαι γκολικός της αριστεράς πρέπει να γνωριστούμε ίσως καλύτερα, αλλά εγώ από 14-15 ετών είμαι ενεργό στην πολιτική και βοήθησα, δεσμεύτηκα τότε για να βοηθήσω ένα εξαιρετικό πολιτικό άντρα, το στρατηγό Ντεγκόλ. Και τότε ε, δεσμεύτηκα για αυτήν την ανθρωπιστική πολιτική. Μπορείτε να την ονομάσετε αριστερά ή δεξιά. Αυτή ήταν η γραμμή μου πάντως. Είναι αυτή η, κοινωνική οικονομία της αγοράς, την οποία μάλιστα διεκδικώ και μάλιστα και κάποιος άλλος ήταν σημαντικός για μένα εκείνη την εποχή. Ο καγκελάριος Αντενάουερ. Αν κοιτάξετε στο γραφείο μου, που είναι ακόμα εδώ στο 13ο όροφο, θα δείτε μια φωτογραφία που μεταφέρω πάντα μαζί μου, που είναι η φωτογραφία του καγκελάριου Αντενάρου για την συνθήκη των Λυσίων και αυτό είναι ο λόγος και της ευρωπαϊκή μου δέσμευση. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία κυρίες και κύριοι για την απέτηση που θα, για να σεβαστώ αυτή, αυτό τον όργο που θα κάνω μπροστά στο δικαστήριο. Είναι πολύ σημαντικό να ορκιστεί κανένας να είναι ανεξάρτητος από όλα τα συμφέροντα και να υπηρετεί το ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτή θα είναι η γραμμή μου για τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Φάπ, σας ευχαριστώ πολύ. Σημειώνω αυτό που λέτε, ότι και με τον τρόπο αυτό θέλετε να συμβάλλετε για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να προσεγγίσει τον πολίτη και προκειμένου να μην προκληθούν μόνο προβλήματα κατά την νομοθετική εφαρμογή, αλλά και πλεονεκτήματα για τον πολίτη. Και ελπίζω ότι η ροζόντια αυτή η εφαρμογή της ε, ενιαίας αγοράς θα διέπεται από τις αρχές που μόλις αναφέρατε. Η εσωτερική αγορά, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου ήδη από τις περασμένες δεκαετίες. Ήδη από την εποχή της ειδικής του άνθρακα ήταν αυτός ο σκοπός. Είναι η κοινή προσπάθεια. Είμαστε μαζί και έχουμε κοινό σκοπό χωρίς να συγχωνευτούμε. Και αυτή η εσωτερική αγορά καλύπτει πολλούς τομείς. Δεν είμαι ο μόνος επίτροπος που είναι ε, με την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς και έχω εδώ τον κατάλογο όλων των επιτρόπων. Νομίζω ότι είναι 13 οι οποίοι λίγο πολύ σχετίζονται με την επιτυχία της εφαρμογής 1.600 νομοθετικών κειμένων που αφορούν την εσωτερική αγορά. Αυτές όμως οι τέσσερις ελευθερίες είναι η καρδιά. Είναι ο σκελετός του ευρωπαϊκού σχεδίου και εγώ θα δεσμεύομαι έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές. Σα ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από την Εύελιν Κεπχάρτ, συντονίστρια από του σοσιαλιστέ. Κυρία Κέπχαρτ, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Μπαρνιέ, να συνεχίσω από εκεί που σταματήσατε. Κατά το παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα τη ενιαίας αγορά, ασκήσε ε, την πολιτική τη αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και την απορρίθμιση. Αυτό ε, εν μέρη με επιτυχία και το Κοινοβούλιο κατάφερε να περάσει επιτυχή σχέδια για, προς το συμφέρον των πολιτών και των εργαζομένων. Και αυτό το είδαμε ιδιαίτερα και στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Το άρθρο 3 το, της Συνθήκης Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ 1η Δεκεμβρίου προβλέπει ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πώς σκοπεύετε να θέσετε με συγκεκριμένα μέτρα αυτή την πολιτική και ποιες πρωτοβουλίες μπορούμε να υπολογίζουμε εκ μέρους σας θα διεξάγετε τακτικά μελέτες κοινωνικού αντικτύπου και θα τις παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Madame εγώ ο ίδιος αναφέρθηκα στην οδηγία υπηρεσίες προηγουμένως και στράφηκα προς εσάς αναφερόμενος και στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να γίνει δυνατή αυτή η οδηγία με βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα είναι δουλειά μου να την καταστήσω εφαρμοστέα ιδιαίτερα για την της, ανθρώπινη της πτυχή. Η ενιαία αγορά λειτουργεί με την αλληλεγγύη και υπενθυμίζω ότι ο Ζακ Ντελόρ πριν από 20 χρόνια όταν ξεκίνησε την ενιαία πράξη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και την βοήθεια του Κοινοβουλίου αμέσως υπέβαλε ένα πακέτο, το πακέτο Ντελόρ για τις πολιτικές συνοχές και αλληλεγγύης τις γνωρίζω αυτές τις ε, πολιτικές γιατί στην προηγούμενη θητεία ως ε, επίτροπος ήμουν επίτροπος για την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική και έτσι καλύπτουμε τα χάσματα ανάμεσα στις περιφέρειες. Θέλω λοιπόν να αναπτύξω ως στρατηγική να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ. Θα το συζητούμε σήμερα αργότερα και μέσω της συζήτησης για τα επαγγελματικά προσέντα, τη δυνατότητα να εγκατασταθεί κανένα σε μια άλλη χώρα, να είναι προστατευμένος όταν κατανολεί, καταναλώνει ιδιαίτερα με ηλεκτρονικές αλλαγές, να έχει ιατρική περίθαλψη σε μια άλλη χώρα, να χρησιμοποιήσει περισσότερα μέσα πληρωμής, να μην έχουμε μόνο δύο κάρτες πληρωμής, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερα προσφορά θέλω να διατηρηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και η καθολική υπηρεσία που προστατεύουν τους πιο απομονωμένους πολίτες εξημών. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, θα υποβάλω μελέτες κοινωνικού αντικτύπου, άλλωστε το επιβάλλει η συνθήκη. Ε, Κυρία Γκέπχαρτ, σας ευχαριστώ. Από την απάντησή σας να συμπεράνω και μπορείτε να μου απαντήσετε αρνητικά ή καταφυτικά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλοι σας το λεπτό, αλλά να θεωρήσω ότι θα ταχθείτε υπέρ μιας κοινωνικής ε, ρήτρας πρόοδου και θα την εντάξετε στην ε, σχετική ρύθμιση για την ιστορική αγορά. Πιστεύω κυρία Γεμπάλ, η απάντησή μου είναι ναι. Εάν πρόκειται για την ρήτρα κοινωνικής κοινωνικού αντικτύπου. Και εγώ προσέθεσα προηγουμένω και περιβαλλοντικού αντικτύπου, αν και δεν προβλέπετε αλλά είναι το ίδιο σημαντικό. Δεσμεύομαι δηλαδή για οποιοδήποτε νομοθετική πράξη θα σα προτείνω, για νέα ή αναθεώρηση, να είναι και αυτή αντικείμενο τη μελέτη αντικτύπου. Και μετά θα πρέπει οι μελέτε αυτέ να είναι ποιοτικέ και θα δούμε το πώ το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα αυτού του αντικτύπου και των μελετών. Για μένα όλα αυτά συμβαδίζουν η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και η κοινωνική πρόοδος συμβαδίζουν. Δεν φαντάζομαι ούτε μία πρωτοβουλία που δεν θα βοηθά την κοινωνική πρόοδο, την πρόοδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η απάντηση είναι καταφατική. Uh, uh Σας ευχαριστώ. Από τη σου ελεύθερος ο ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενη Επίτροπε, μια εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χρήζει μια αποτελεσματικής εφαρμογής που δεν θα ορθώνει ε, κολλήματα περιτά στους ε, καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από αυτό το πρίσμα η εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας είναι κρίσιμη, γιατί η εναρμόνιση είναι μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία και πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην ενσωμάτωση των κοινωτικών οδηγιών στην εσωτερική νομιτάξη. τάξη. Και κάθε χρονιά όταν εξετάζουμε τους διάφορες πίνακες ε, εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί τόσο ε, εύρυθμα και απρόσκοπτα όσο θα επιθυμούσαμε. Ποια είναι τα μέτρα που έχετε στη στο μυαλό σας για να διευκολύνετε την διαδικασία της εναρμόνισης. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε λιγότερη νομοθεσία αλλά πιο αποτελεσματική, χρησιμοποιώντας κανονισμούς ως νομοθετικό εργαλείο και όχι οδηγίες. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας αυτόματος και συστηματικός κανόνας που συνηγορεί υπέρ της χρήσης του κανονισμού από της οδηγίας εξαρτάται από τις ε, περιστάσεις. Άλλοτε είναι δόκιμη η διοδική και άλλοτε ο κανονισμός. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και τα εργαλεία που μας δίνει το εφνομοθετήν, δηλαδή και τις μελέτες επιπτώσεων και τις ε, νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη, κυρία Γκέπχαρτ, και όπως είπα είναι πολύ σημαντικές. Κοινωνική επίπτωση, περιβαλλοντική επίπτωση. Στη συνέχεια θα καταρτήσουμε σχέδια οδηγιών, σχέδια κανονισμών και όσοι βρίσκονται εκτός του Κοινοβουλίου και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να μάθουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση τον τομέα του ανταγωνισμού, δεν αποφασίζει, προτείνει και άλλοι αποφασίζουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των πολιτών και το Συμβούλιο των Υπουργών είναι οι συνομοθέτες και αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις. Θέλουμε φυσικά να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και σωστά η κοινοτική νομοθεσία και θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ε, κάποια εξουσία και καταστολή δηλαδή διαδικασίες επί και επιβολή κυρώσεων και θα δείξουμε πυγμή, θα είμαστε αυστηροί, θα ζητήσουμε πειθαρχία, αλλά θα προτιμούσα πριν φτάσουμε στην καταστολή να προσπαθήσουμε με πειθό, με διάλογο, συστηματικό διάλογο να πείσουμε τα κράτη-μέλη. Έχουμε ενδιαφέρουσε διαδικασίε όπω το Solvit που αρχίζει και λειτουργεί σωστά ή το EU Pilot για τα προβλήματα με τι χώρες. Και πολύ συχνά θα μεταβαίνω επί τόπου. Δεν πρόκειται να μείνω χειρωμένο στο γραφείο μου στι Βρυξέλλες. Δεν θα μείνω στο γραφείο μου. Μία φορά την εβδομάδα θα πηγαίνω σε μία κοινοτική χώρα και δεν θα πηγαίνω μόνο στις πρωτεύουσε, θα επισκέπτομαι και τις περιφέρειες. Θα επιστρέψω και στις περιφέρειες, γιατί ως αρμόδιος για τις περιφέρειες επίτροπος, για την περιφερειακή πολιτική, πήγαινα πολύ συχνά. Και θα συν... συνεργαστώ με όσους φορείς μπορούν να με βοηθήσουν για να εφαρμόζουμε σωστά την κοινωτική νομοθεσία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε το παράδειγμα δύο οδηγιών που αναφέρατε και εσείς, την οδηγία για τις υπηρεσίες και την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και εκεί υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Αναφέρατε το Solvit. Είμαι ο εισηγητής ε, της ε, Επιτροπής για το Solvit. Πολύ καλό μέσο το Solvit για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επιλύσουν διάφορα προβλήματα. Αλλά το Solvit δεν, μπορεί, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τη χρήση της διαδικασίας επί παραβάση, για παράδειγμα. Ερωτώ λοιπόν, θα δράσετε με πυγμή και θα υιοθετήσετε κάποια στεναρά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσετε την σωστή και άμεση μετάθεση της κοινοτική νομοθεσίας σε περίπτωση που κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Κύριε Μπούζοη, η απάντησή μου είναι καταφατική. Δεν θα ήθελα να κάνω δική προθέσεων όμως εδώ. Σίγουρα Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εμπόδισαν ε, τη σωστή εφαρμογή των δύο οδηγιών σε πολλά κρατημέλη, τι οδηγίε για τι υπηρεσίε και για τα επαγγελματικά προσόντα, και θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί. Μέχρι τα τέλη του έτους σας υπόσχομαι ότι θα μεταβώ προσωπικά στις 27 χώρες μέλη και θα έχω ημερήσεις συναντήσεις με όλους εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με το θέμα αυτό. Φυσικά πρώτα με τους υπουργούς γιατί δεν μπορώ να δράσω ερήμη των αρμόδιων υπουργών, αλλά θα συναντηθώ και με διοικητικούς υπαλλήλου και με οικονομικούς και οικονομικούς εταίρους που ασχολούνται με την εφαρμογή. Και θα πάω και πιο μακριά, αλλά πρώτα θέλω με τα μάτια μου να διαπιστώσω πού βρίσκεται το πρόβλημα πριν αναλάβω δράση. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Χάιντι Ρούλε από τους Πράσινους EFA. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαρνιέ, ο κύριος Μπαρόσο δήλωσε ότι θα κάνει θα αναλάβει πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ως προς το περιβάλλον. Εσείς θα είστε υπεύθυνο για την ιστορική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, τι θεωρείτε ότι περιλαμβάνει ε, ο τομέας των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, για παράδειγμα την παροχή υδατός. Θα προσπαθήσετε να ενοποιήσετε την αγορά και τι σκοπεύετε να κάνετε σε ό,τι αφορά και την ε, οδηγία για τα ύδατα. Μιλάτε για μια νομοθετική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά της ε, παροχή υπηρεσιών. Θα υπαχθεί και σε αυτό η οδηγία για τα ύδατα. Και ενδεχομένως να υπάρξει και σχετική οδηγία. Πώς θέλετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε στο θέμα της παροχής υπηρεσιών τις μεγάλες παραδόσεις και τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στις παραδόσεις σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Κυρία Ρούλε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδική νομοθεσία για τις, εταιρικές, για τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ε, ιδιωτικού φορέα ή τις παραχωρήσεις. Για τα απορρίμματα, την επεξεργασία των αποβλήτων και τους βιολογικούς καθορισμούς, Έχουμε τέτοιες ε, συμπράξεις ε, κράτους και ιδιωτών ή υποχωρήσεις ό,τι αφορά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, υπάρχει ανακοίνωση για την ανάγκη ανάπτυξης τέτοιων συμπράξεων ε, μεταξύ κράτους και ιδιωτικών φορέων. Είναι εταιρικέ σχέσεις όμως, εταιρικέ συμπράξεις και μάλιστα τέτοιου είδους θέματα καλύπτονται από ένα τμήμα των νομοθεσιών για τις κρατικές προμήθειες, αλλά η παραχώρηση υπηρεσιών δεν καλύπτονται από νομοθετικά κείμενα. Ο ρόλος μας είναι να μην αφήσουμε τις επιχειρήσεις ή ε, τοπική αυτοδιοίκηση σε μια κατάσταση ανασφάλειας δικαίου μέσα στην εσωτερική αγορά. Θα τα σκεφτώ λοιπόν όλα αυτά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη, κυρία Ρούλε, αν χρειάζεται μια νέα οδηγία για το θέμα αυτό. Θα δούμε αν είναι σκόπιμο να προτείνουμε μια νέα οδηγία. Και θα μεριμνήσω πρώτα απ' όλα, όπως προτείνατε κι εσείς, να λάβω υπόψη όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, τις παραδόσεις ε, για τα θέματα αυτά των παραχωρήσεων σε όλα τα κράτη-μέλη, στις περιφέρειες, ακόμη και στα γερμανικά κρατήδια. Ξέρω ότι εργάζεστε με ζέση και εκπονείτε μια συνολική έκθεση απολογισμού για την εσωτερική αγορά και σίγουρα και η δική σας έκθεση θα μας χρησιμεύσει στην επεξεργασία αυτού του θέματος. Σα ευχαριστώ και θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Δυστυχώ δεν απαντήσατε όμω τι θα κάνετε για τα ύδατα. Αν θα κάνετε κάτι θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό. Κατά δεύτερον να σα ευχαριστήσω για τι επεξηγήσει σα σε ό,τι αφορά για τι παραχωρήσει. Ε, υπηρεσίων. Νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού με την Επιτροπή το Κοινοβούλιο να βρει λύσεις, γιατί είμαι υπεύθυνη για μια έκθεση σε ό,τι αφορά τέτοιες ε, αναθέσεις έργων και βλέπω ότι υπάρχει ε, μεγάλη γραφειοκρατία και πολλές κοινότητες, πολλοί δήμοι ε, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και για εξωτερικές παροχές, για εξωτερικές συμβουλές, το οποίο είναι πάρα πολύ επίπονο. Είναι το αντίθετο αυτό που θέλουμε να πατήχουμε με την καλή νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Όλοι γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του ύδατος και της ανάγκης ε, ποιοτικού ύδατος, ακόμη και στη δική μας Ήπειρο, που νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στο απειρόβλητο των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Τις προάλλες, στη Νότια Γαλλία, ε, η εποχή του τρίγου μέσα σε 20 χρόνια έχει γίνει τρεις ε, εβδομάδες νωρίτερα. Έχει μετατοπιστεί πολύ νωρίτερα. Οπότε όλα τα θέματα διαχείρισης ύδατος και ποιότητας ύδατος είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, υπάρχουν ε, διαφορετικές υπηρεσίες ύδατος στην Ευρώπη και όλα τα θέματα του ύδατος θα καλυφθούν από ένα γενικό κείμενο και για τις αναθέσεις έργου και για τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Τώρα, γιατί θα πρέπει το είδωρο να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από τις αναθέσεις ή το θέμα των απορριμμάτων και της εξυγένσης. Αυτά θα τα συζητήσουμε όλα αργότερα μαζί. Uh, uh thank you for that. ευχαριστώ από την ομάδα ECR, ο κ. Αταμπίλαν. Ευχαριστώ. Ένα τμήμα των ερωτήσεων που ήθελα να σας υποβάλω το έθιξαν οι συναδέλφοι. Οπότε θα ήθελα να σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο θέμα, την... Ε, ένα κανονισμό που λήγει στα τέλη του Μαΐου Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε νέο κανονισμό που παρά τις προηγούμενες δηλώσεις ε, ε, παραλείπει κατά τη γνώμη μου σημαντικά θέματα για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Για παράδειγμα, παραλήφθηκε το πολύ σημαντικό άρθρο 4 του προηγούμενου κανονισμού για την πρόσβαση ανεξάρτητων εργαστηρίων σε τεχνικές πληροφορίες, ε, διαγνωστικού εξοπλισμού ή προγραμματισμού. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το θέμα των διατάξεων για τα, τους χονδρέμπορους και τις, τους διανομής αυτοκινήτων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί θεμητός ανταγωνισμός, κάτι που επηρεάζει την, το εύρος επιλογής των καταναλωτών αλλά και το ύψος των τιμών. Τι διαβήματα ε, θα κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, εκατομμυρίων ε, καταναλωτών που διαθέτουν γιοταχή. <laughs> Είπατε να προστατεύσετε τους καταναλωτές, τους ευρωβουλευτές. Δεν νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές χρήζουν προστασίας. Uh, Σίγουρα και οι ευρωβουλευτές οδηγούν ή κάποιοι οδηγοί είναι και ευρωβουλευτές. Ε, κύριε Μπιέλα, θα εξετάσω την ερώτησή σας. Φαντάζομαι ότι μιλήσατε όχι μόνο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας γιατί υπάρχουν πάρα πολλά διασυνοριακά προβλήματα σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και, και εσείς επισημάνατε πολλές αδυναμίες για το εμπόριο αυτό. Δεν ξέρω αν αναφερόσταν μόνο στην αυτοβιομηχανία ή καλύπτεται και άλλους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων. Θέλω περισσότερο χρόνο για να ετοιμάσω, την απάντηση. Φαντάζομαι το κατανοείτε. Να σας βοηθήσω γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μπίλεν αναφερόταν ε, σε θέματα τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και διαστάσεις που αφορούν τους καταναλωτές. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει μία επερώτηση ο κύριος Μπίλαν ή μήπως να περάσω στον επόμενο ομιλητή. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Κυρίως ε, αφορά στις αμπλόκ ε, εξαιρέσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και το ε, σχέδιο BR 2010 που περιλαμβάνει κάποιες οδηγίες που είναι πολύ ανακριβείς στη διατύπωσή τους. Δεν έχουν μόνο σήμαντη ερμηνεία και πολύ συχνά μπορεί να δημιουργηθούν παρερμηνίες ή να χρησιμοποιηθούν από ε, ομίλους ε, αυτοκινήτων εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ανακρίβεια αυτών των διατάξεων ίσως αποβεί εις βάρος των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την επιλογή τους και το, τις τιμές των αυτοκινήτων, γιατί θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις ε, μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων. Αυτό ζήτησα από τον Επίτροπο να εξετάσει. Κύριε Μπιέλαν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, σίγουρα οι εξαιρέσεις που αναφέρατε αφορούν πολλούς τομείς. Μερικοί εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων μου. Θα το εξετάσω όταν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Θα αναλύσω αυτό το ειδικό θέμα που θίξατε για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά υπάρχει άλλος αρμόδιος επίτροπος για τις επιχειρήσεις. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν για, τα... για την οδηγία και τις υπηρεσίες είναι αυτό το θέμα των εξαιρέσεων. καλό είναι όταν εφαρμόζεται μια οδηγία να μην υπάρχουν μαζικές εξαιρέσεις. Και δεν είναι αυτό απλό το θέμα. Θα πρέπει να αναλυθεί κατά περίπτωση κάθε εξαίρεση. Θα κάνω μια ενδελεχή εξέταση μετά από διάλογο με τις διαφερόμενες χώρες και το ώστε να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί αυτός ο αριθμός των εξαιρέσεων. Σας ευχαριστώ που διευκρινίσατε το ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ο κύριος Κυριάκος Τροντεφλίτης εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, η αξιολόγηση της εσωτερικής αγοράς ε, εξακολουθεί να γίνεται βάσει κριτηρίων που δείχνουν την κινητικότητα των υπηρεσιών του κεφαλαίου και των εργαζομένων. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Ε, στην δική μας προσέγγιση ως ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά ε, θεωρούμε ότι κεντρικό στοιχείο είναι ο άνθρωπος, όχι η επιχείρηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να διευκρινίσετε συγκεκριμένους κοινωνικούς όρους τους οποίους σκοπεύετε να επιδιώξετε για να πετύχετε τους φιλόδοξους στόχους που έχετε θέσει. Ε, ε, ε, Κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως είπα πριν από λίγο στην κυρία Γκέπχαρτ ή και στον κύριο Σβάμπ, για μένα είναι αδιανόητη η πρόοδος της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη πρόοδο. Φυσικά υπάρχει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών αφενό και επιχειρήσεων αφετέρου. Η επιχείρηση είναι ένα τόπο παραγωγή που στηρίζεται στην τεχνογνωσία, στι δεξιότητε, στην ευφία των ανδρών και των γυναικών. Και χρειαζόμαστε όλε τι επιχειρήσει ε, και τι μικρέ και τι μεσαίε και από από τα 5 εκατομμύρια επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη, το 90% είναι μικρές ε, έως και πολύ μικρές που, εργα... που λειτουργούν με έναν έως πέντε εργαζόμενους. Οπότε ισχύει η ίδια απάντηση που έδωσα προηγουμένως. Θα προσπαθήσω να δώσω αυτή την ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση στην εσωτερική αγορά. Θα επεξεργαστώ συγκεκριμένα σχέδια για την ε, εγκατάσταση των ανδρών και των γυναικών, την προστασία των κοινοφελών υπηρεσιών, την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πριν από λίγο αναφέρθηκα σε μια άλλη ιδέα που μου είναι προσφυλής, για επικερδείς επιχειρήσεις μεν, προσοδοφόρες, αλλά ταυτόχρονα για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα αναλάβω κι εγώ για να επαναφέρω μια κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση στην πολιτική της εσωτερικής αγοράς. Εκτός μικροφώνου. I'm sorry. I repeat. Επαναλαμβάνω, η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας έχει θέσει ένα νέο πλαίσιο για τις κοινωνικές πτυχές της ενιαίας αγοράς. Πώς θεωρείτε ότι η νέα συνθήκη θα επηρεάσει τις ε, αποφάσεις σε θέματα όπως Λαβάλ και Βίκιν. Η συνθήκη της Λισαβόνας για την οποία έδωσα μάχη όπως και πολλοί από εσά. Για πολλούς τομείς ε, κατοχυρώνει τη διαδικασία της συναπόφασης, παρόλο που ίσχυε ήδη για τις περισσότερες ε, αρμοδιότητες ε, του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς. Και εισάγει την οριζόντια κοινωνική ρήτρα, την ανάγκη εκπόνηση μελέτη κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτέ οι νέε ρήτρε για μένα δεν είναι απλώ τυπικό θέμα. Είναι πολύ ουσιαστικό και θα συνεργαστούμε στενά και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να εντατικοποιήσουμε αυτό το διάλογο, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να καταρτήσουμε ποιοτικού νόμους και οδηγίες. Πριν από λίγο αναφέρθηκα σε άλλα θέματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν ε, ε, το αντικείμενο ε, νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους μικροαποταμιευτές, προτα... προτάσεις για να καταπολεμηθούν τα τοκογλυφικά επιτόκια, ενιαίος τρόπος πληρωμών, εμπορικός τομέας. Όλα αυτά τα θέματα αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και εμπίπτουν και στην εσωτερική αγορά. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε τον γύρο των συντονιστών, ο κύριος Σαλβίνη από την ομάδα EFD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ που έρχομαι από τη Σαββοία, με άκουσα ιδιαίτερα τα όσα είπατε για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά της των απομιμήσεων. Θέλω να μου πείτε πότε, πώς με τι κόστος, σε πόσους μήνες, γιατί εγώ προέρχομαι από την Βόρεια Ιταλία, από την Παδανία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα από τις απομιμήσεις. Και ρωτώ λοιπόν, κυρία Μελλοντική Επίτροπε, πώς προτίθεστε να προστατεύσετε την παραγωγή, την πνευματική ιδιοκτησία και πώς θα εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές τι καταναλώνουν, από πού προέρχονται, το, τι τρώνε, το τι, πού προέρχεται ο, ο υπολογιστής που χρησιμοποιούν. Γενικά πιστεύω ότι ο καταναλωτής αγοράζει τρόφιμα φυσικά για τη διατροφή του, αγοράζει φάρμακα για την ίασή του και δικαιούται να γνωρίζει την προέλευση αυτών των προϊόντων, πώς παρασκευάστηκαν, πώς παρήχθησαν, αν οι παραγωγοί τους ε, σέβονται τους ε, κανόνες και τις προδιαγραφές. Πολλές φορές πρόκειται και εισαγόμενα προϊόντα και εκεί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα της συχνηλασιμότητας και το απέδειξα όταν ε, είχα αναλάβει τον αγροπιστιστικό κλάδο στη χώρα μου. Όχι για λόγους προστατευτισμού, αλλά για λόγους προστασίας, για την εξασφάλιση του θεμητού ανταγωνισμού. Εγώ είμαι υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά υπέρ του θεμητού ανταγωνισμού. Είναι λογικό να προστατεύουμε τους καταναλωτές σε θέματα υγείας και διατροφής. Επισημάνεται τις απομιμήσεις. Υπολογίζονται σε 2,5 εκατομμύρια η απόλυτο θέσεων εργασίας εξαιτίας αυτού του φαινομένου, της μάστιγας των απομιμήσεων, με τους κινδύνους που ανέφερε και για την ανθρώπινη υγεία και τον σφετερισμό των ε, σημάτων, ε, των εμπορικών σημάτων και των, ε, των δικών μας μαρκών. Θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια λοιπόν να προστατεύσουμε αυτά τα εμπορικά μας σήματα, τις μάρκες μας, τις παραδόσεις που κατέληξαν στην παραγωγή τους. Γι' αυτό, αυτό θα συνεχίσω τη στενή συνεργασία με τους συναδέλφους Ντεγκούχτ, τα Γιάννη, ώστε και τα θέματα ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης που είναι αρκετά καθόδη και η εμπορική συμφωνία κατά των απομιμήσεων που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επιμερίσουμε καλύτερα το, την προσπάθεια καταπολέμησης α, παγκοσμίως των απομιμήσεων και των προϊόντων πειρατείας. Σας ευχαριστώ και βεβαίως έχετε κατά ότι το Μιλάνο είναι μια βόρεια πόλη που θα ήθελε πολύ να είναι έδρα του παρατηρητήου γιατί είμαστε και οι δήμονες σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Από δική μου πλευρά λοιπόν έχετε υποστήριξη στη δραστηριότητά σας για αυτό το μέτωπο. Καλό θα ήταν και ο τομέας των ειδών διατροφή να γίνει πιο επαγγελματικός και εντός της εσωτερικής αγοράς και Υπάρχουν διαφορές και στις δεξιότητες ανάλογα και με τα διπλώματα, που εκδίδονται στην Ευρώπη. Ο οδηγό τυρ είναι διαφορετικό, σε διαφορετικό δίπλωμα αυτό που λαμβάνει στην Ιταλία ή στη Βρετανία. Ε, και ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εναρμόνιση που θα έπρεπε να εξετάσει και αυτή η Επιτροπή. Δεν πρόκειται τώρα να σχολιάσω αυτά που είπατε για τους ε, ε, δασκάλους του σκι. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά το θέμα δεν είναι να ε, εμποδίσουμε έναν Άγγλο, Ρουμάνο, Γάλλο δάσκαλο σκι ή οδηγονταλίκας να ασκήσει αλλού τη δραστηριότητα. Το θέμα είναι η ασφάλεια όμως. Ένας δάσκαλος σκι ή ένας οδηγός βαρέου οχήματος θα πρέπει να ασκησει αλλο τη δραστηριοτητα το θεμα ειναι η ασφαλεια ομως ενας δασκαλος δεξιότητες είναι τεράστιο το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, πάντως θα φροντίσω να εξασφαλιστεί ένας συντονισμός, μία σύγκληση, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Επίσης, για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απομίμησης και Πειρατείας, θα πρέπει να συγκεντρώνει στοιχεία και για τις κοινωνικές επιπτώσεις, ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας για να λάβουμε αντίστοιχη δράση και αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής ε, Ιστορικής Αγοράς. Η πρώτη ερώτηση από την κυρία Ρόζα Τούνφουν του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, η εμπειρία σας από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσήλωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ιδέα και το κουράγιο σας είναι γνωστά της πάση. Και Όλοι βλέπουμε τις πρόοδους της εσωτερικής αγοράς, αλλά οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν απολαμβάνουν εμπράκτος πολλές φορές τις ευκαιρίες που τους δίνει η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε βελτιώσεις και στην ενημέρωση. Είπατε ότι είστε πρόθυμος και ανοιχτό στο διάλογο, όχι μόνο στις πρωτεύουσες, αλλά και σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Το θέμα της συνεργασίας ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών αρχών ε, χρήζει βελτίωσης. Μιλούμε για τον κοινωνικό αντίκτυπο, για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αλλά αρκούν όλα αυτά. Προτίθεστε να ε, προτείνετε στο Σώμα των Επιτρόπων ε, τη λιδία λίθο της εσωτερικής αγοράς ώστε να μην υπονομευθεί η εσωτερική αγορά από τις υπόλοιπες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τέσσερις ελευθερίες που ανέφερα προηγουμένως, που είναι η ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού σχεδίου και εμπίπτει στι αρμοδιότητε δικέ μου και άλλων περίπου δέκα επιτρόπων, ο σεβασμό αυτών των τεσσάρων ελευθεριών και η έμπρεκτη εφαρμογή του, κυρία Βαντούν, είναι πραγματικά η λιδία στο του έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν χρειάζεται να το υποβάλω αυτό το τεστ, αυτή τη δοκιμασία στου επιτρόπους. Υπάρχει αυτή η οριζόντια κοινωνική ρήτρα που ανέφερα και οι βασικέ αρχέ τη εσωτερική αγορά θα πρέπει να τηρούνται από όλου του επιτρόπους, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ έχω περισσότερε αρμοδιότητε για να εξασφαλίσω την εφαρμογή του, αλλά οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση περνάει και από το τεστ, από τη δοκιμασία τη εσωτερική αγορά. Γνωρίζουμε ότι ο κατακαιρματισμός αυτής της αγοράς ε, αποτελεί ένα πρόβλημα και εμείς θα είμαστε θεματοφύλακες αυτής της εσωτερικής αγοράς, αλλά και σκαπανείς. Και θα, δεν θα αφιστώ προσπαθειών και ενέργειας προκειμένου να πείσω τους συνομιλητές μου και να τους κάνουν να αντιληφθούν τη σημασία της σωστής εφαρμογής. Μία ιδέα που, μας, που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι να συναντώ τακτικά τους αρμόδιους με την εφαρμογή των κειμένων της εσωτερικής αγοράς, ώστε να γίνεται μια ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, μια κοινωνία ιδεών και μια καλύτερη και πιο αποτελεσματικότερη συνεργασία. In order to... Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά, θα πρέπει να εμπλακούν και τα συμφέροντα των ε, εμπλεκομένων φορέων για να είναι πιο συγκεκριμένες οι δεσμεύσεις τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Άρα, για το μέτρο αυτό που μόλις ε, αναφέρατε, έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την υποστήριξη του προγράμματος του Φόρουμ της Εσωτερικής Αγοράς, το οποίο έχουμε συζητήσει εδώ, στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Κύριε το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία και αυτό είναι ο μύτος της αριάδινης ε, της συμπεριφοράς μου, αν ε, επικοινωθώ ως Επίτροπος. Θέλω να φέρω τους ανθρώπους κοντά για να καθίσουμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας και να αποφασίσουμε τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσουμε μέσω οδηγιών, κανονισμών και προπολογισμού. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Εσωτερική Αγοράς ε, είναι πολύ καλή ένα τέτοιο ευρωπαϊκό φόρουμ ε, θα φέρνει κοντά εκπροσώπους των εθνικών φόρουμ. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως, γιατί είναι υπερβολικός ο κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς. Το λέω χαμογελώντας, αλλά την την εποχή του δημοψηφίσματος ακούσατε το ποταπό επιχείρημα για τον Πολωνό Ιδραυλικό. και αν μιλήσουμε για ένα Λουξεμβούργιο Ιδραυλικό. Δεν είμαι καθόλου περήφανος για όλη αυτή την ε, επιχειρηματολογία και την αντιπαράθεση. αντιπαράθεση. Ένας Λουξεμβούργιος ε, για να κινηθεί 30 χιλιόμετρα χρειάζεται να, χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τέσσερα διαφορετικά διοικητικά έγγραφα. Αυτή τη γραφειοκρατία θα πρέπει να καταπολεμήσουμε που είναι δαπανηρή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μειώθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύριο το διοικητικό κόστος με κάποια μικρή απλούστευση. Θα ήθελα στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να μειώσουμε κατά 7 δισεκατομμύρια τις δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χάρη στην ελάφρυνση της γραφειοκρατίας που θα προτείνουμε. Σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Μπερναντέ Βερνιό, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής από τους Σοσιαλδημοκράτες. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, το θέμα της προστασίας αποτελεσματικών και ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών είναι βασικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς και της εδαφικής ακαιρεότητας. Η συνθήκη της Λισαβόνας λαμβάνει καλύτερα υπόψη αυτές τις υπηρεσίες. Όμως, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην ενσωμάτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες απαιτούν διευκρίνηση. Λυπάμαι λοιπόν εδώ που η επιστολή για την θα καθήκοντά σας δεν αφέρει καθόλου σε αυτά τα θέματα ούτε και στις γραπτές σας απαντήσεις. Όμως ο πρόεδρος Μπαρόζο δεσμεύτηκε το Σεπτέμβριο και παραθέτω εδώ να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, πράγμα το οποίο θα δείξει τη σημασία του στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Δεσμεύεστε να προτείνετε μια οδηγία πλαίσιο για τις κρατικές υπηρεσίες και αν ναι, πότε και εγγράφομαι πλήρω στο σχέδιο που παρουσίασε ο Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο, που αναφέρθηκε σε ένα πλαίσιο ποιότητα για τι κρατικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία και πριν να θέσετε το ερώτημα, στα εισαγωγικά μου σχόλια, και λυπάμαι που δεν το έγραψα στις γραπτές μου απαντήσεις, γιατί αν τα είχα γράψει όλα εκεί δεν θα είχατε ερωτήματα να μου θέσετε σήμερα. Οπότε καλύτερα να συμπληρώσουμε σε αυτές τις τρεις ώρες ακρόασης και τις γραπτές απαντάσεις που σας έθεσα. Αλλά για μένα είναι προφανές, είναι τμήμα αυτής της ασάφειας που πρέπει να εξαφανιστεί για την Ευρώπη και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ξέρω ποια είναι η ανησυχία και μετά την οδηγία για τις υπηρεσίες για την καλή εφαρμογή των κοινωνικών δημοσίων υπηρεσιών. Υπάρχουν υπηρεσίες πολύ σημαντικές για τους πολίτες που αποκλείονται, όπως η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας ε, δημοσίου συμφέροντος. Αλλά θέλουμε να πάμε ακόμα παραπέρα. Αυτή είναι η ιδέα μου, να μην υπάρχουν πλέον καθόλου ασάφειες με ένα καλό κείμενο. Εσείς το ονομάζετε οδηγία πλαίσιο. Υπάρχουν όμως και πολλές παραδόσεις, πολύ διαφορετικές ανάλογα με τις χώρες και τις ίδιες τις περιφέρειες. Τώρα χρειάζεται οδηγία πλαίσιο, χρειάζεται οδηγία ανατομέα και το λέω αυτό γιατί στην Επιτροπή πρώτη έγινε αυτή η συζήτηση και μεταξύ συναδέλφων που ήταν σοσιαλιστές και είναι πάντα. Δεν ήταν αναγκαστικά ξεκάθαρο ότι για να εξασφαλίσουμε αυτήν την εγγύηση των κρατικών υπηρεσιών και δημοσίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα άτομα, χρειάζεται αναγκαστικά ένα γενικότερο πλαίσιο και όχι τομεακές οδηγίες. Αλλά είμαι ανοιχτό, δεν κλείνω την πόρτα, αυτό μπορώ να σας πω. Σα ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Έχω κάποιες δυσκολίες με αυτό το, την ονομασία πλαίσιο ποιότητα. Είναι πολύ ασαφές. Καταλαβαίνω τι εννοείτε, αλλά σήμερα μπορείτε να μας πείτε αν θα προτείνετε ένα νομοθετικό ή νομικό εργαλείο για αυτές τις υπηρεσίες που είναι σημαντικές και τις αναφέρατε την υγεία και πρέπει να βοηθήσουμε και τους ηλικιωμένους και τους ανήλικους. Είμαστε μια ήπειρος η οποία γυράσκει και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Απάντηση οι υπηρεσίε τις οποίες αναφερθήκατε, η υγεία είναι από τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα και ηλικιωμένα άτομα ή τα πιο απομονωμένα άτομα, αποκλείονται από τα υφιστάμενα κείμενα και με αυτή τη λογική προστατεύονται. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κάποια αμφιβολία και εγώ θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να συνεργαστούμε για να μην υπάρχει πλέον αυτή η ασάφεια. Δεν είναι ρόλος της Κομισιόν ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμποδίσει με βάση την πολιτική ανταγωνισμού τέτοιου είδους υπηρεσίες να προσφερθούν επί τόπου όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός με άλλη χώρα. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, γιατί και αυτό περιμένετε ίσως, ακόμα και αν ένας επίτροπος δίνει στο κολέγιο των επιτρόπων την προσωπική του, την προσωπική του άποψη. Αλλά στην απάντησή σας ήδη αναφερθήκατε σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Χρειάζεται πλαίσιο γενικό ή διαφορετικό πλαίσιο για κάθε μία από αυτές τους τομείς. Ε, δεν είμαι σίγουρος για το ποια είναι η απάντηση αυτή τη στιγμή. Θα εργαστώ πάντως με τη λογική που σας περιέγραψα. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Καλνιέτη από την ομάδα του ΕΛΚ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, πριν μπω στην πολιτική ήμουν στα δημιουργικά επαγγέλματα δραστήρια και ξέρω το πόσο η πειρατεία είναι σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη και είναι εμπόδιο στη δημιουργικότητα. Πολλά κράτη-μέλη ανέλαβαν πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, οι οποίες όμως δεν βαίνουν όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν θα ήταν σκόπιμο να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καθορίσουμε ένα κοινό νομικό πλαίσιο κατά πολέμηση των απομνημίσεων και της πειρατείας για να έχουμε μια πραγματική ενιαία αγορά δημιουργικού περιεχομένου. Euh, είναι βασικό θέμα. Σας είπα ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων απασχόλησεων που έχουν εξαφανιστεί εξαιτία αυτής της ε, απομίμησης και της ε, πειρατείας. Είναι εκθετική η αύξηση της κατάστασης και η σοβαρότητα της κατάστασης με βάση την παγκοσμιοποίηση και ρωτάτε αν χρειάζεται ένα διαφορετικό ή νέο πλαίσιο. Έχω εδώ ένα κατάλογο όλων των ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων για την απομίμηση και τις παραχαράξεις από το 2004 ακόμα και από το 1977 για τα σήματα. Έχουμε ένα σωρό κείμενα και εγώ πριν κάνω ένα νέο κείμενο θα ήθελα να ελέγξω την αποτελεσματικότητα αυτών των υφιστάμενων κειμένων. Υπάρχουν 179 εκατομμύρια προϊόντα τα οποία κατάσχονται στα σύνορα το 2008. Το 2007 ήταν πολύ λιγότερα, υπήρχε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση και θα χρησιμοποιήσω όλες τις δυνατότητες δράσης που έχουμε και τις εργασίες του νέου παρατηρητηρίου και το φόρουμ για να μας βοηθήσουν να υιοθετήσουμε τα σωστά μέτρα για να είμαστε αποτελεσματικοί μόνοι μας εδώ στην Ευρώπη αλλά και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Και να πω δύο λόγια μετά το ερώτημά σας για την πειρατεία μέσω του ίντερνετ. Όλοι από την παιδική μας ηλικία ε, έχουμε μια κάποια αδυναμία για τους πειρατές. Για την πειρατεία όχι όμως. Ε, εγώ θα δεσμευτώ για τα δημιουργικά επαγγέλματα και στο ίντερνετ πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα. Υπάρχει βεβαίως η ελευθερία ενημέρωσης και πληροφόρησης, αλλά πρέπει να αποζημιώσουμε και τους δημιουργούς και δεν μιλάμε μόνο για τους μουσικούς και πρέπει να αποθαρρύνουμε τη δημιουργία που είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Μαζί με την κυρία Ρέντινγκ λοιπόν και άλλους συναδέλφους θα συνεργαστούμε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία πληροφόρησης και ενημέρωσης και προστασία των καλλιτεχνών. Μιλήσατε για τις απομιμήσεις. Το παρατηρητήριο κατά των απομιμήσεων που ιδρύθηκε τον Άνοιξη του 2009 έχει σκοπό να μαζέψει τις απαραίτητες πληροφορίες για υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία στην εσωτερική αγορά. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δομή αυτού του παρατηρητηρίου έτσι ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικό ποια είναι τα σχέδιά σας στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Γενικά πιστεύω ότι για να δράσουμε σωστά πρέπει να κατανοήσουμε σωστά. Και γενικά θα ήθελα αντικειμενικές και αμερόληπτες παρατηρήσεις για να καθοδηγήσουμε τις εργασίες της Κομισιόν των συνεργαστών και η νομοθετική προσπάθεια να βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Είπατε και εσείς η ίδια ότι το παρατηρητήριο δεν είναι και πολύ ηλικιωμένο, μόλις ξεκίνησε τις εργασίες του. Θα δώσει κάποια στοιχεία για τις ε, ε, επιπτώσεις των αποσμιμήσεων και ε, θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε κοινέ εκστρατείε για την ευαισθητοποίηση του, της κοινή γνώμης και να προχωρήσουμε και σε πιο ξεκάθαρες θέσεις νομοθετικού περιεχομένου, προτάσεις και μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση διεθνώς για αυτή την Διεθνή Εμπορική Συμφωνία. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν θα καταπολεμήσουμε τις απομιμήσεις χωρίς να έχουν οι άλλες περιοχές του κόσμου τις ίδιες απαιτήσει, γιατί από εκεί προέρχονται πολλά από τα προϊόντα που είναι αντικείμενο των απομιμήσεων. Σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Μπάρμπαρα Βέιλερ από τους Σοσιαλδημοκράτες για την επόμενη ερώτηση. Κύριε Μπαρνιέ, εγώ εδώ είμαι, εδώ είμαι. Να επανέλθω στο θέμα της κοινωνικής πτυχής της εσωτερικής αγοράς. Θα έχετε διαπιστώσει σίγουρα ότι τα πολλά ερωτήματα που έχουν τεθεί για το θέμα αυτό καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας. Και σας λέω ότι οι απαντήσεις σας ως τώρα μου δείχνουν ότι και εσείς το παίρνετε πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό, πιο πολύ στα σοβαρά από ότι προκατοχό σα. Θέλω να σα ρωτήσω όμω συγκεκριμένα πώ θα διευκρινίσετε τη θέση σας με τα κράτη-μέλη, όχι με εμάς, εμείς στην πλευρά, μας, στην πλευρά σας είμαστε, για να τεθούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, περιβαλλοντικά κριτήρια και να εφαρμοστούν τα κριτήρια αυτά. Αν τα συστήσουμε τα κριτήρια αυτά, αν τα απαιτήσουμε, πώς θα ξεκαθαρίσετε στα κράτη-μέλη ότι η απλοποίηση και ότι η μείωση της γραφειοκρατίας δεν σημαίνουν αυτόματα την απορρίθμιση και πώς θα ξεκαθαρίσετε και στα κράτη-μέλη γιατί αυτό το βλέπουμε καθημερινά ότι οι υπηρεσίες για την κοινωνική πρόνοια δεν θα πρέπει να περάσουν αυτόματα στον ιδιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είστε σίγουροι ότι θα ξοδέψω πολύ χρόνο και ενέργεια για να εξηγήσω ότι δεν είναι η Κομισιόν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που παρεμποδίζει την ιδιωτικοποίηση της μίας ή της άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Θα εξηγήσω τι απαιτείται σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, να εξηγήσω τα κείμενα για την ενιαία αγορά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά τίποτα παραπάνω. Δεν θα αναλάβουν οι Βρυξέλλες, εμείς όλοι, τα όσα γίνονται με βάση την επικουρικότητα και την κυριαρχία των κρατών μελών και των περιφερειών και την πολιτική βούληση των μεν και των δε. Γι' αυτό θα είμαι ξεκάθαρος. Τώρα, ας περάσουμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τις κρατικές προμήθειες θα χρησιμοποιήσω τα, τις κρατικές προμήθειες. Είναι 2-3 ευρώ για να κάνουμε ό,τι λέει η συνθήκη. Δηλαδή να ενισχύσουμε την δημόσια δράση των τοπικών αρχών για να λάβουν καλύτερα στις εργασίες τους αυτές τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις και ακόμα και για την έρευνα και την καινοτομία. Είμαι πεπισμένο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ του ε, τους κρατικούς διαγωνισμούς και τις κρατικές προμήθειες. Εγώ για 17 χρόνια ήμουν τοπικά εκλεγμένος άρχοντας και ήμουν ένας από τους πρώτους πρόεδρους που εισήγαγε το 1% των κρατικών προμηθειών για το περιβάλλον. Είχαμε μια χάρτα και υποχρέασαμε την ε, ε, τοπική μας κυβέρνηση για τα οδικά έργα να βάλουν μια υποχρεωτική ρήτρα για χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων στην προσφορά που έκαναν. Κατασκευή οδών παραδείγματος χάρων. Ε, αντί να πάρουμε μια πρώτη ύλη στη φύση, μπορούμε να ανακυκλώσουμε ε, καταδεφασμένα κτίρια για να έχουμε χαλίκι. Στην την Γαλλία υπάρχουν 7.000 επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν έτσι τα υλικά και θα ήθελα αυτή η πρακτική να γενικευθεί και αυτό θα το κάνουμε μέσω των κρατικών προμηθειών. Και έχω την πρόθεση να συνεργαστώ ιδιαίτερα με την Επιτροπή των Περιφερειών και τις τοπικές αρχές. Δεν θέλουμε να τα επιβάλλουμε από πάνω προς τα κάτω, αλλά να συνεργαστούμε με τις περιφέρειες για να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Βάιλερ ε, δεν θα θέσει δεύτερη ερώτηση και να περάσω στον κύριο Ζουβά, ο οποίος θα θέσει το επόμενο ερώτημα. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, στην πολιτική σας καριέρα πάντα ήσασταν υπέρ της Ευρώπης της άμυνας και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης ε, είχατε προεδεύσει και στην γέννηση της Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού και ένας από τους ρόλους της είναι να δημιουργήσει ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνιστική του αμυντικού εξοπλισμού. Όμως αυτή η αγορά είναι πολύ κατακαιρματισμένη. Οι κρατικές αγορές αμυντικού εξοπλισμού ε, είναι πολύ ε, εθνική και αυτό απορρέει ότι υπάρχουν εμπόδια σε όλη την αμυντική αγορά. Αυτό είναι εις βάρος της ε, ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανία και ε, επιβάλλει ένα μεγάλο βάρος στα δημόσια οικονομικά. Οπότε ρωτώ, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα έχετε προτάσεις να μας υποβάλλετε για να ε, διορθωθεί η κατάσταση. Απάντηση. Είπα και εξ αρχής ότι είμαι εδώ μπροστά σας ως πολιτικός άνδρας και είμαι πεπισμένος ότι πέρα τα όσα πρέπει να κάνουμε για την αγορά θα πρέπει η Ευρώπη να έχει μια πολιτική διάσταση. Αυτό περιμένουν και οι πολίτες άλλωστε και τα όσα γίνονται στον κόσμο, ένας ασταθής άδικος και ευάλωτος κόσμος, επικίνδυνος κόσμος δείχνει ότι πρέπει να δώσουμε στην Ευρώπη μια δυνατότητα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής πριν να πάμε, όπως λέει και η συνθήκη, προς την ευρωπαϊκή άμυνα. Το θέμα αυτό δεν έχει προχωρήσει πολύ και αυτό γιατί αγγίζει την καρδιά της εθνικής κυριαρχίας. Φύγουμε πολύ λεπτά θέματα και δικαιολογημένα άλλωστε γιατί ε, ε, θίγουν το απόρριτο των προμηθειών ή την εμπιστευτικότητα και όλα αυτά προστατεύονται από τα 3, 346 άρθρο της συνθήκης και ε, κράτη-μέλη το χρησιμοποίησαν πολύ αυτό το άρθρο για να μην υπάρχει κοινή χρήση αυτών των εξοπλισμών. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι και σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε άλλους, η κοινή χρήση είναι το κλειδί. Θα έχουμε μια καλύτερη άμυνα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα έρευνας, τους εξοπλισμούς. Αυτό κάνει και ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός που θα προεδρεύσει και η συνάδελφός μου κυρία Άστον. Στο δικό μου τομέα και εδώ εκφράζομαι πλέον ως Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά έχουμε μια οδηγία η οποία δεν είναι και πολύ παλιά την οποία όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ενσωματώσουν, που όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ενσωματώσουν μέχρι το 2011, που λαμβάνει υπόψη την ευαίσθητο χαρακτήρα αυτού του τομέα και θα πρέπει να προαγάγει την κοινή χρήση στον τομέα αυτό. Θα δώσω λοιπόν κάθε στήριξη και θα χρησιμοποιήσω την πειθώ γιατί θέλω να συνεισφέρω για μια ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική έτσι ώστε και η Ευρώπη και τα λέω εδώ σοβαρά δεν είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε πάντα υπεργολάβοι υπεργολάβοι της αμερικανικής οικονομίας ή της κινέζικης οικονομίας δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα υπό επιρροή αυτό απαιτεί όμως αμυντική πολιτική και εξωτερική πολιτική οπότε θα συνεισφύρω φέρω και εγώ για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αγορά αμυντικού εξοπλισμού Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, αλλά για να επανέλθουμε σε αυτόν τον περίεργο χαρακτήρα αυτής της αγοράς που είναι και εξαιρετικός και οι αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης είναι 170 δις ευρώ με 80 δις ως αγορές υπάρχει αυτή η έννοια των αντισταθμιστικών ωφελών που είναι ότι ε, ο αγοραστής απαιτεί αντισταθμιστικά ωφέλη για τις εθνικές του επιχειρήσεις Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ιστορικές συνήθειες, αλλά το ερώτημα είναι πιστεύετε ότι αυτές οι πρακτικές, οι συνήθειες συνάδουν με ένα μοντέρνο κοινοτικό δίκαιο. Απάντηση. Δεν θα προχωρήσουμε ποτέ κατά των κρατών μελών και μειώνοντας την κυρίαρχή τους θέση στον τομέα αυτό. Μαζί τους μόνο και η αναγκαιότητα επίσης θα μας οδηγήσει στον τομέα και τα όσα γίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα ενθαρρύνουν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να οικοδομήσουν αυτήν την κοινή άμυνα. Αναφερθήκατε σε αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Είναι πολύ συγκεκριμένη παράδοση που υπάρχει στις αμυντικές αγορές. Εγώ αντικειμενικά, και αυτή είναι η πεποίθηση μου, αυτές οι πρακτικές είναι αντίθετες με την συνθήκη και οδηγούν σε διακρίσεις. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον ανταγωνισμό για αυτές τις κρατικές προμήθειες. Νομίζω λοιπόν ότι χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο χρόνο για να εξηγήσουμε και ε, ελπίζοντας ότι όλη η οδηγία αυτή για την άμυνα θα σωστή, σωστά θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη, νομίζουμε ότι θα πετύχουμε να περατωθεί πλέον αυτή η πρακτική. Κύριος Ρόσφορ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που αναφέρατε και το οποίο είναι κάτι κυρίως απασχολεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και 30 χρόνια και αφορά πολλούς εξημών εδώ. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και επίγει το να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό γιατί αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση που γνωρίζουμε. Πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε όλη την δημιουργικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι τα πραγματικά θύματα από την απουσία αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο ευρωπαϊκό. Τον περασμένο χρόνο είχαμε ένα σημαντικό βήμα γιατί έχουμε ε, πλέον τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρωτεχνία και έχει πλέον το, ε, καθιστά το ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο. Ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε ότι πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα τώρα από εδώ και πέρα. Και η θέση σε ισχύ του ευρωπαϊκού αυτού διπλώματος εξαρτάται από την υιοθέτηση του κανονισμού που διαχωρίζει το θέμα του γλωσσικού καθεστώτος. Τι θα κάνετε εσείς, Λίαν, συντόμως για το θέμα αυτό. Απάντηση. Μιλήσαμε για την ισχύ, την κυριαρχία της Ευρώπης, τη δυνατότητα να μην είναι σε υπεργολαβία και την ισχύ της οικονομίας. Αυτό το θέμα διαρκεί πολύ καιρό και δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και για να δώσω συνέχεια στα όσα είπε ο κύριος Ροσφόρ, ένα δίπλωμα που καταθέτει μια επιχείρηση για 13 13 κράτη-μέλη κοστίζει 10 φορές παραπάνω από ό,τι στις ΗΠΑ. 20.000 ευρώ για να καταθέτει καθένας κάποιος προστασία σε 13 κράτη-μέλη και όχι στα 27. Σας έφερα εδώ γυαλιά. Δεν είναι τα δικά μου που κατασκεύασε μια επιχείρηση στη Βενετία. Είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα φημισμένο στις ΗΠΑ. Η επιχείρηση που το κατασκευάζει αυτό δεν μπόρεσε να καταθέσει δίπλωμα ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη. Γιατί κοστίζει πολύ ακριβά. Οπότε προστατεύεται στι ΗΠΑ και σιγά σιγά έτσι χάνουμε την οικονομική μας ισχύ. Χαίρομαι και εγώ λοιπόν όπως και εσείς που υπήρξε αυτό το πρώτο βήμα στο Συμβούλιο Υπουργών. Κύριε με αυτή τη συμφωνία πριν τα Χριστούγεννα για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία, που αυτή τη στιγμή αποκλείει το θέμα του γλωσσικού καθεστώτο, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Ξέρω ότι η Ισπανική Προεδρία με την οποία θα συνεργαστούμε θέλει να προωθήσει το θέμα και για το γλωσσικό θέμα θα ήθελα να προτείνω λίγαν συντόμω ένα κανονισμό κύριε Ροσφόρ. Θέλω να χρησιμοποιήσω τι τεχνολογικέ προόδου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αυτόματη μετάφραση για να πείσω τα κράτη-μέλη που δεν είναι ακόμα πεπισμένα ότι πρέπει να βρούμε το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και υπάρχει και το θέμα της δικαιοδοσίας επίσης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνοδεύσουμε αυτό το νέο σύστημα του ευρωπαϊκού διπλωμάτου ευρωδιεθνούς με ένα ειδικό ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα αυτά τα διπλώματα που να καλύπτει και τη δική μας επικράτεια αλλά και άλλες χώρες γιατί αυτό αφορά και την Ελβετία παραδείγματο χάρη. Κύριος Ροσφόρ, συνεχίζω την ερώτησή μου για το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων τεχνίων, το οποίο λίγο πολύ, ακόμα και αν δεν λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά, κάπως λειτουργεί. Όμως με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και της αναγνώρισης αυτής της οντότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικό πρόσωπο, υπάρχει η δυνατότητα η Ένωση να προσχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίων, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε και την προσχώρηση του συνόλου της επικράτειας της Ένωσης σε αυτό το θεσμό και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αυτού του βήματος και της Ένωσης και να έχουμε συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Είστε υπέρ αυτής της προσχώρησης της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο διπλωμάτων ευρεία Απάντηση ναι, αν αυτό επιλύσει το πρόβλημα. Αλλά εσεί έχετε μεγαλύτερη εμπειρία για το θέμα και εγώ θα βασιστώ στην απόψη σα. Αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα νομικώ πώ. Ξέρω τι κάνει και το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Υπάρχουν 600 άτομα που εργάζονται εκεί, αλλά είναι πολύ περίπλοκο νομικά το θέμα από ό,τι το περιγράφεται. Ε, μου λένε πάντως ότι μια προσχώρηση στη σύμβαση απαιτεί αρμοδιότητα της Ένωσης και είναι για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλετε θα ήταν πιο εύκολο προηγουμένως να έχουμε συμφωνήσει για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Τεχνίας Θα ήθελα από κοινού να έχουμε μια απόφαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Τεχνίας και από ό,τι μου λένε οι νομικοί μετά μόνο από αυτή τη συμφωνία θα έχουμε μία ευκαιρία να γίνει αυτή η προσχώρηση στη σύμβαση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ευχαριστώ και νομίζω ότι έχω... Είμαι πολύ ενεκτικό γιατί έχουμε άλλου τρει ε, ομιλητέ και ξέρω ότι έχω και του συναδέλφου που θα ακολουθήσουν. Μία ερώτηση λοιπόν για του τρει επόμενου ομιλητέ για να συντομεύσουμε. Η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι η κυρία Επίτροπε. Ελπίζω αυτή τη φορά να ακούσετε καλά τη διερμηνία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε ο καλεσμένος σημερινής ακρόασης και έχω να ρωτήσω το εξή. Είπατε ότι σας είναι προσφυλές το θέμα της αναθέρμανσης της εσωτερικής αγοράς και χαίρομαι ιδιαίτερος. Με ενδιαφέρει όμως ιδιαίτερα η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Γιατί το δυναμικό αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τεράστιο για την οικονομική επιτυχία της Ευρώπης. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που αισθάνονται στο πετσί τους ε, τα προβλήματα από το κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Κατά τη γνώμη σα, ε, τι τομεί τη εσωτερική αγορά θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να υποφεληθούν καλύτερα από ε, τι ευκαιρίε τη εσωτερική αγορά και τι πρωτοβουλίε θα αναλάβετε ως αρμόδιος επίτροπος για την εσωτερική αγορά προκειμένου να ευνοήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Euh, Σα ευχαριστώ κύριε Χάντζλικ. Σας ευχαριστώ που χύσατε λίγο φως σε αυτό το θέμα. Σας είπα ότι η προτεραιότητά μου είναι η αναθέρμανση της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να την ε, ξανεστανθούν δικοί τους οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί λέμε ότι ευνοούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 70% δηλαδή των ευρωπαϊκών θέσεων απασχόλησης. Ένα από τους, στόχου ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας Εφνομοθετήν είναι να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις για τις α, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξοικονομήσουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, πέραν ε, των προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό είναι και ο στόχο του Small Business Act, ε, τη νομοθετική πράξη του Ιουνίου του 2008 για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και θα είναι θέματα και του δικού μου χαρτοφυλακίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία του Small Business Act. Η γενίκευση του τεστ των μικρών επιχειρήσεων, η απλούστευση σε ό,τι αφορά τη χορήγηση κάποιων ενισχύσεων, κώδικα ε, καλών πρακτικών για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει ένα θέμα που το γνωρίζει ο πρόεδρο Λένε, γιατί αφοσιώθηκε ψυχείται και σώματι στο θέμα αυτό και είναι το θέμα τη ε, Ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία, γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το, καταστατικό αυτό τη ε, ευρωπαϊκή Εταιρείας. Όλε αυτέ είναι προσπάθειε που στόχο έχουν να διευκολύνουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ε, θέλουμε να μειώσουμε και το κόστο κάποιων νομικών υποχρεώσεων για τη δημοσίευση των λογαριασμών του, για παράδειγμα. Επίσης υπάρχει το θέμα της ενιαίας θηρίδας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε αυτή την ενιαία θηρίδα. Δεν ξέρω αν θα είναι μία αναχώρα ή ανα, αναπεριφέρεια. Εδώ σέβομαι την επικουρικότητα, αλλά θέλω η ενιαία θηρίδα να λειτουργήσει για να μην χρειάζεται να παραπέουν μεταξύ 10 διαφορετικών διοικήσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για τις διατυπώσεις τους. Ο καθηγητής ε, Κορέαντε Ντεκάμπος έχει το λόγο τώρα από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κύριε Επιτροπέ, κύριε Μπαρνιά, εδώ είμαι. Δεν αφιβάλλουμε για την ικανότητά σας και την, το ενδιαφέρον σας και την προθυμία σας να επισκεφτείτε χώρες και περιοχές. Θυμόμαστε την επίσκεψή σας μιας φτωχής κοινότητας στο Ράβο Πέισε, στις Αζόρες και μάλιστα έχουμε πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από την επίσκεψη εκείνη. Βέβαια, από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, διαπιστώνω ότι η οδηγία και τις υπηρεσίες δεν είναι καλό παράδειγμα στις εταιρικές αγοράς, γιατί είπατε ότι λυπάστε ε, για, την, για τον κατακαιρματισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ 13 επιτρόπων. Οπότε, για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, θα, θα ζητήσετε τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο του κατακαιρματισμού σε μια τόσο ε, πολυπρόσωπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προσέκρουσε στην απροθυμία πολλών κρατών μερών. Πώ αντιδράσετε, θα προωθήσετε την αναθεώρησή της, θα πιέσετε τις χώρες να τη δεχτούν ή θα, θα προτείνετε μια έκθεση μελέτη επιπτώσεων ή αξιολόγηση. Κύριε Κορέρα Δεκάμπος, ούτε και εγώ έχω ξεχάσει την επίσκεψή μου στις Αζόρες. Και αν μου δείξετε την εμπιστοσύνη σας, θα φροντίσω ο Αρμόδιος Επίτροπος να ασχοληθεί με τις 7 υπεραπόμακρες περιοχές. Να μην τις ξεχνούμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει το παρόν σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου να μην ξεχάσει αυτές τις υπεραπόμακρες περιοχές. Και εξακολουθώ να είμαι αφοσιωμένος στις δεσμεύσεις μου για τις υπεραπόμακρες περιοχές. Η Επιτροπή είναι ένα σώμα διαφορετικό από τις κυβερνήσεις. 13 επίτροποι είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των 1.600 νομοθετικών κειμένων που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Και θα ε, εργαστούμε συλλογικά. Κάθε επίτροπος έχει το επιτελείο του, έχει το γραφείο του και παρακολουθεί και αυτά που κάνουν οι συνάδελφοί του. Και εγώ θα είμαι... θα επαγρυπνώ για την σωστή εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου. Αναφερθήκαμε σε δύο οδηγίε προηγουμένω για τι υπηρεσίε και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία για υπηρεσία έχει ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέτε ότι αντιβαίνει στην εσωτερική αγορά. Αν δεν την εφαρμόσουμε ή αν την εφαρμόσουμε πλημελώ. Αν την εφαρμόσουμε σωστά όμω, εξασφαλίζοντα τα απαραίτητα εχέγγυα για τι κοινοφελεί υπηρεσίε, η οδηγία για τι υπηρεσίε δεν αντιβαίνει στην εσωτερική αγορά. Είναι θετική αρκεί να εφαρμοστεί σωστά. Γι' αυτό και η προσωπική μου προσπάθεια είναι να πείσω τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν σωστά αυτές τις οδηγίες και να τις αξιολογήσουν. Είμαι υπέρ της αξιολόγησης όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και θα μεταβώ, όπως σας είπα, προσωπικά σε κάθε χώρα για να το φροντίσω. Τελευταίος ομιλητής από τους πράσινους, ο κύριος Καμφά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρνιέ. μας μιλήσατε για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τις ε, προθέσεις σας. Μπορείτε να αναλάβετε εδώ και τώρα δέσμευση ενώπιόν μας να μην ε, ε προτείνετε εφαρμογή της χώρας προέλευση στη θητεία σας αν αποβεί αρνητική για τους εργαζόμενους. Μπορείτε να δεσμευθείτε απέναντι στους επιτρόπους ε, και να υποβάλλετε αξιολόγηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους που έχει επισύρει σωρία κριτικών από τα συνδικάτα. Ποια είναι η ανάλυση σας για, τα, για τις αποφάσεις του ΔΕΚ, Λαβάλ, Βίκιν και άλλες. Συμφωνείτε με την ομολογία του ΔΕΚ ή θα προτείνετε άλλες πρωτοβουλίες ε, για διαφορετική ερμηνεία του δικαίου. Μπαρνιέ. Φυσικά είμαι ανοιχτός, έτοιμος και πρόθυμος, όπως είπα και προηγουμένως, για να προβώ σε μια αντικειμενική αξιολόγηση των κειμένων, των νομοθετικών κειμένων. Θα ήθελα και μια αντικειμενική αξιολόγηση τη οδηγία για τους αποσπασμένους. Αυτό δεν με ρωτήσατε. Λέω ναι στην αξιολόγηση. Α μην ξαναρχίσουμε μια παλιά συζήτηση για τη χώρα προέλευση. Θυμάμαι πολύ καλά αυτό το θέμα και ήδη από την αρχή της ομιλία μου και στάθμισα πολύ σοβαρά τα λόγια μου, δεν έχω καμία πρόθεση να κυλιδώσω το όνομά μου και τα καθήκοντά μου με απόπειρα επιδείνωσης της κοινωνικής κατάστασης. Θέλω η εσωτερική αγορά να γίνει εργαλείο για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη. Υπάρχει νομολογία του 10 και δεν την παραμερίζουμε ούτε την αγνοούμε. Θα την αξιολογήσουμε, θα την εκτιμήσουμε και πριν γίνει μια σωστή αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν θα υποβληθεί καμία περαιτέρω πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την ε, τις πολύ συνεκτικές του απαντήσεις και σας ευχαριστώ και εσάς συνάδελφοι που ήσασταν συνοπτικοί. Να καλέσω τον κύριο Μπαρνιέ να κάνει ένα πολύ σύντομο τελικό σχόλιο, όχι παραπάνω από ένα λεπτό, αν θα θέλετε να κάνετε μια τελική παρατήρηση. Δεν είχα προβλέψει να μακρηγορήσω γιατί ήδη ξεπεράσαμε το χρόνο του πρώτου τμήματος της ακρόασης και έχουμε φάει λίγο από το χρόνο της δεύτερης ακρόασης, του δεύτερου τμήματος. Ολοκληρώνω λοιπόν το πρώτο τμήμα με κάτι που είπε και στην αρχή. Θα ήθελα να επαναφέρω τους άνδρες και τις γυναίκες στην καρδιά της πρότασης ε, και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Εσωτερική Αγορά. Το είπα και προηγουμένω για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να εξυπηρετεί του άνδρε και τι γυναίκε και όχι το αντίθετο. Αυτή είναι η δική μου ακράδαντη πεποίθηση. Και αυτό θα το επιχειρήσω σε σχέση και σε συνεργασία με το περιβάλλον που είναι ένα λίκνο ευαισθησιών, δεξιοτήτων, εμπειριών και τεχνογνωσίες και έχω ήδη περάσει πολλούς επικοδομητικούς και ενδιαφέροντες μήνες εδώ από την ε, θητεία μου ως Ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, όχι με νοσταλγία, αλλά με ευχάριστες αναμνήσεις, γιατί δεν κάνουμε πολιτική με νοσταλγική διάθεση, αλλά είχα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα πάρει την Προεδρία η κυρία Μπόουλς για το δεύτερο ήμιση της ε, ακρόασης. Okay, everybody. Um, Να ξεκινήσουμε και σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως, γιατί έχουμε καθυστερήσει και λίγο. Να ευχαριστήσω τον Μάλκομ που λίγο συντόμευσε τους ομιλητές τους τελευταίους. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς ε, Έχουμε λίγη έλλειψη χρόνου και θα περιορίσω λίγα δευτερόλεπτα τον χρόνο ομιλία των συναδέλφων. Κύριε Μπαρνιέ, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, σας καλωσορίζω σας, παρακαλώ. Μην κάνετε φασαρία, μόνο εγώ μιλάω τώρα. Κύριε Μπαρνιέ, σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Αναφερθήκατε στα εισαγωγικά σας σχόλια στην κόποση... Και όπως ξέρετε, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν υπάρχει περιθώριο για κόπωση. Έχουμε υποσχέσεις του G20, ρήτρες αναθεώρησης, περίπου 50 νομοθετικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κατά πάσα πιθανότητα είναι διπλάσιος αριθμό αν προσθέσουμε και την επιτροπολογία. Πρωτού σας δώσω τον λόγο για τα εισαγωγικά σας σχόλια, θα ήθελα να θέσω τρία σημεία τα οποία ελπίζω ότι μέχρι το τέλος θα μπορέσετε να μου απαντήσετε καταφατικά. Καταρχάς, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τρεις αρμόδιοι επίτροποι για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, χρηματοπιστωτικές αγορές και ανταγωνισμό, θα πρέπει να συνεργαστούν στενά. Και θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για όλους αυτούς τους τομείς της πολιτικής και θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη συνένωση των πολιτικών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε να δεσμευτείτε εσείς προσωπικά για ένα σύστημα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την Επιτροπή μας στον τομέα αυτό που άπτεται πολλών χαρτοφυλακίων. Κατά δεύτερο, στην ερώτηση σας απάντηση είπατε ότι θα κάνετε μελέτες αντικτύπου. Συμφωνείτε να αναλύσετε επίσης και το σωρευτικό αντίκτυπο της, ε, του προγράμματος νομοθεσίας μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Και κατά τρίτον, θα ήθελα να τονίσω, γιατί αναφέρατε στη γραπτή σας ε, απάντηση, ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τους ε, βουλευτές, με τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό θα σήμαινε πιο πολύ διάδραση. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι δύσκολο σε ό,τι αφορά και τον όγκο της δουλειάς που έχουμε, αλλά και το, την πίεση, την χρονική που προέρχεται από το G20. Προτείνουμε λοιπόν να συμμετέχει το Κοινοβούλιο πιο πολύ στην ε, προκαταρτική, ανεπίσημη φάση και αυτό θα εξίσωνε αν θέλετε και το ρόλο του Κοινοβουλίου με το ρόλο των εμπειρογνωμόνων. Αυτό σας το αναφέρω ως μία σκέψη. Και ελπίζω να έχετε να καταφέρετε να θυμηθείτε τα σχόλια αυτά μέχρι το τέλος. Πέντε λεπτά για τα εισαγωγικά σας σχόλια προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Και όπως ξέρετε, ξέρω πώς να κλείσω το μικρόφωνο γιατί έχω το κουμπί off. Οπότε σας δίνω το λόγο. Chair, uh, for giving the floor. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Όπως είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει δρεωμένη εσωτερική αγορά χωρίς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η κόπωση εδώ δεν χωρά. Διανύουμε την σοβαρότερη οικονομική χρήση από το 1929. Χωρίς μια άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πολιτικών και νομισματικών αρχών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα αντιμετωπίσουμε μια σωρία χρεοκοπιών και θα επισέλθουμε σε μια ε, σοβαρότερη κρίση εμπιστοσύνη και πιο μακροχρόνια ύφεση. Η κρίση έχει κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες ε, και συνεπιφέρει και άλλες κρίσεις όπως την επισητιστική ε, που επηρεάζει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο και δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις. Ξέρω ότι αυτά ανησυχούν και εσάς. Και γι' αυτό δημιουργήσατε και άλλωστε μια ειδική τέτοια επιτροπή για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Όπως ε, κυρίες και κύριε, κυρία Πρόεδρος είπε, ο, το αρχικό σχόλιο του Πίτσπερκ, πρέπει να ξεκινήσουμε μια εποχή ευθύνης. Θα πρέπει η διαφάνεια, η ευθύνη και η ηθική να τοποθετηθούν στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η κρίση ήταν πολύ σοβαρή. Ας μην ε, υποκρινόμαστε ότι πρόκειται να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις. Καμία αγορά, κανένας φορέας, κανένα προϊόν, καμία περιοχή δεν θα πρέπει να ξεφύγει πλέον από τις ε, σχετικές νομοθεσίες και από την αποδοτική εποπτεία. Το ίδιο έθεσε και ως απέτηση η Άγγελα Μέρκελ πριν από κάποιες εβδο, ε, εβδομάδες. Θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις του G20 και η Ευρώπη είναι δεσμευμένη για τη διαδικασία αυτή σε παγκόσμια κλίμακα και θα πρέπει η Ευρώπη να είναι παγκόσμια τέτοια κινητήριος δύναμη. Από την ίδια αποφασιστικότητα περιμένουμε και από τους εταίρους μας πέρα από το G20 θα αφιερώσω χρόνο και ενέργεια για διμερείς σχέσεις αποτελεσματικές με τους βασικούς μας εταίρους. Αυτός είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κυρίε και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει επίση να φέρουμε ει αίσιο πέρα ε, τη μεταρρύθμιση τη εποπτεία, ώστε να γίνουμε η πρώτη περιοχή του κόσμου που θα αντλήσει διδάγματα από την κρίση αυτή. Θα ήθελα να ότι φόρο τιμή στο αξιέπαινο έργο του Ζακ Ντελαροζιέρ και του επιτελείου του και θα ε, μείνουμε πιστοί στο έργο αυτό με τον συνάδελφο Λιρέν. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η σωστή προσέγγιση για την ρύθμιση των εναλλακτικών ταμείων και θα υποβάλω προτάσεις για τους κανόνες ε, φερικιότητας των τραπεζών και για το επίπεδο ε, και την ποιότητα του επίπεδου του κεφαλαίου τους. Επίσης θα υποβάλω νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα παράγωγα προϊόντα και το, την ενίσχυση των ε, επιμελητηρίων ψήφισης. Επίσης θα επανεξετάσω εις βάθος την οδηγία για την, κατάχρηση των αγορών και δεν θα φύγω τα καθόδη ζητήματα όπως είναι οι κυρώσεις ή οι ακάλυπτες πωλήσει. Είναι τομεί όπου δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω. Φερεγγιότητα 2, αναθεώρηση της οδηγίας MIFID, λογιστικά πρότυπα και προληπτικά πρότυπα, ε, συντάξεις, όλα αυτά τα θέματα θα τα εξετάσω υπό το φως των εργαλείων του εφνομοθετή. Ε, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Η οικονομία μας χρειάζεται ε, ρύθμιση και ανάλογη με τις αγοράς. Επίσης, ε, έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις ε, σε παιδίσεις, ασφαλίσεις. Ε, θέλουμε καινοτόμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η χρηματοπιστωτική μας αγορά θα γίνει πιο ανταγωνιστική αν έχουμε καλούς κανόνες που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Η Ήπειρός μας με τα πλεονεκτήματα που έχει θα έχει και η φόρο πλεονέκτημα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αν καταφέρει να υιοθετήσει μία αποτελεσματική και ευφυή ρυθμίση που θα ε, εξασφαλίζει μια σταθερότητα η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει μόνο με υγιεί χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε που θα βρίσκονται στην υπηρεσία τη οικονομία και όχι το αντίθετο. Αυτό είναι μία από τι απαραίτητε προποθέσει για να οικειοποιηθεί ε, και πάλι ο πολίτη ε, την εσωτερική αγορά και τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Σα προτείνω λοιπόν να συνεργαστούμε προκειμένου ο χρηματοπιστωτικό μα κλάδο να γίνει καλύτερα ρυθμιζόμενο και αποτελεσματικό. Επίση, θέλω πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με ένα υγιές, ανοιχτό και υφόρο περιβάλλον και θα ήθελα να συνεργαστούμε για να εξετάσουμε θέματα που αφορούν τον καταναλωτή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εγγύηση των αποταμιεύσεων, τα ενυπόθηκα δάνεια και ευρύτερη επιλογή χαρτών, καρτών για τους καταναλωτές. Και πιστεύω ότι θα βγούμε από την κρίση όχι όπως μπήκαμε. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματά μας και να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε και αυτό το εργοτάξιο θέλω να το ανοίξουμε από κοινού. Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο και να εφοδιαστούμε με εργαλεία για να, να προβλέψουμε, να προλάβουμε και να διαχειριστούμε μελλοντικές κρίσεις. Γι' Αυτέ είναι οι σκέψεις μου, κυρίε και κύριοι. Αντί να εξοδεύουμε ενέργεια και χρήμα για να διορθώνουμε τις προηγούμενες κρίσεις, καλύτερα να επενδύσουμε στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής οικονομίας με πράσινη ανάπτυξη, την σταθερότητα, την ειρήνη στον κόσμο, την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την ε, καταπολέμηση των δημογραφικών προκλήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω πολύ για να μην σας πάρω το χρόνο και να περάσουμε κατευθείαν στον πρώτο γύρο ερωτήσεων ο Ζαν Πολ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενο Επίτροπε, ως συντονιστής του ΕΛΚ έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να ανοίξω το πυρ των ερωτήσεων. Μέσω του καταλόγου που μας απαριθμίσατε, μας υπενθυμίσατε πόσο η Επιτροπή είναι προσιλωμένη σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί πριν ακόμη ξεσπάσει η κρίση, η Επιτροπή μα είχε επισημάνει την ανάγκη δράση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ ε, έπεσε σε ότα κοφώνει η προειδοποίησή μα. Πάντω, ε, βλέπουμε την αποφασιστικότητά σα ε, για πολλά από τα θέματα αυτά. Πώς θα λάβετε υπόψη τι ανησυχίε και τον προβληματισμό τη οικονομική μα επιτροπή για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Γκοζές για, για τα λόγια σας. Φυσικά θα συνεργαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη και για κείμενα για τα οποία επεξεργάζεται όπως τα hedge funds ή το θέμα της εποπτείας και πολλά άλλα ζητήματα με τα οποία θα συνεχίσω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσχετα με το τι έκανε η απερχόμενη Επιτροπή. Για όλα αυτά τα θέματα θα στηριχθώ στην τεχνογνωσία της ε, Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων. Είστε πραγματικά ένα φυτόριο απόψεων, ε, ευφυΐας, πραγματογνωμοσύνης και πολλοί έχετε εμπειρία από επιχειρήσεις, από τράπεζες, Είστε οι δήμονες. Ένας επίτροπος δεν είναι παντογνώστης, μπορεί να έχει πεπιθήσεις, αλλά δεν είναι γνώστης των πάντων. Γι' αυτό και επικουρείται ε, από ένα επιτελείο ειδικών. Ο κύριος Κουίστον Ντέβιτ Ράιντ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, θα με βοηθήσουν. Θα στηριχθώ λοιπόν και στη δική σας ε, γνώση και εμπειρία ώστε όπως πρότεινε και η κυρία Σαρον να καταρτήσουμε ποιοτικέ νομοθετικές διατάξεις, καλούς νόμους και μην αφιβάλλετε ότι θα είμαι κοντά σας όποτε το ζητήσετε ώστε να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το πνεύμα κατά την ε, έναρξη των καθηκόντων. Είναι τεράστιο αυτό το έργο που έχουμε να πραγματοποιήσουμε. Είναι ένα ογκώδες νομοθετικό πακέτο και αυτό που υπάρχει τώρα και αυτό που θα υποβληθεί στο μέλλον και θα ήθελα να προβώ σε μια πλήρη και διεξοδική αξιολόγηση αυτού του νομοθετικού πακέτου. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην οικονομική χρησιμότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συμφωνούμε. Είστε έτοιμος να πάτε ακόμη πιο μακριά. Ε, τι γίνεται με την κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες, γιατί και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πού στηρίζεται η κερδοσκοπία που διαπιστώνουμε εδώ και δύο-τρία χρόνια, που είναι ένα καινούριο φαινόμενο στις πρώτες ύλες. Δεν μιλώ για την ενέργεια, ε, το πετρέλαιο κτλ. Αν αποδείξουμε κερδοσκοπία ε, τέτοιου είδους ε, για, τα, για τις γεωργικές πρωτεσίλες πραγματικά είναι σκανδαλώδη. Σας είπα ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από την πείνα, λιμοκτονούν. Ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, στην Αϊτή για παράδειγμα, κύριε Κοζές, είναι χώρα μάρτυρας και υποφέρει τα πάνδυνα η Αϊτή. Πριν από ένα χρόνο, τη στιγμή, την εποχή του λοιμού, βλέπαμε γυναίκες στο Πόρτο Πρά στην Αϊτή να δίνουν στα παιδιά τους να τρώνε μπισκότα λάσπης με λίγο λάδι από πάνω. Είναι απαράδεκτο αυτό ε, για πολιτικούς ηθήνοντες ε, αυτό το θέαμα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τα παράγωγα προϊόντα γιατί με αυτά συνδυάζεται η κερδοσκοπία για τις πρώτες ύλες και σίγουρα θα μεριμνήσουμε να αποκαταστήσουμε μια διαφάνεια και έναν έλεγχο αυτών των κερδοσκοπικών τάσεων στις πρώτες ύλε μέσω των παράγων προϊόντων. Ο κ. Μπούλμαν από τους Δημοκρατές. Κύριε Μπαρνιέ, και εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, της Επιτροπής σας ορίζουμε εδώ στην ακρόαση αυτή. Αναφέρεται ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κινητήριος δύναμη και λέτε επίσης ότι θα πρέπει όχι μόνο να επανορθώνει και να κάνει επισκευές, αλλά εξ αρχής να δώσει νέα κατεύθυνση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα ήθελαμε να ακούσουμε πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου για την ηθική σας ε, ε, διάθεση, αλλά πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να ε, θυσιάσουμε το βραχυπρόθεσμο, το μακροπρόθεσμο μάλλον μέλλον των αγορών με βραχυπρόθεσμα κέρδη. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτά. Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε τη μακροπρόθεσμη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Κύριε Μπούλμαν, Σίγουρα δεν στερούμε βούλησης, θέλησης για δράση και σας ε, διαβεβαιώνω ότι στάθμισα πολύ σοβαρά τα λόγια μου. Υπάρχει δέσμευση για να προχωρήσω και, θα... και νομίζω ότι έχω χαίρο της εμπιστοσύνης ε, και της υποστήριξης και του κυρίου Μπαρόζο αλλά και του κυρίου Ρεν και του συναδέλφου Αλμούνια και άλλων επιτρόπων φαντάζομαι γιατί θα συνεργαστώ με πολλούς για όλα αυτά τα θέματα θα αντιλήσουμε πολλά διδάγματα και ένα από αυτά, από τις νομοθετικές προτάσεις, είναι θα πρέπει να κατανοήσουμε για να δράσουμε πρώτα και να δράσουμε στο σωστό επίπεδο με αποτελεσματικά εργαλεία εποπτείας και τον απαραίτητο παγκόσμιο συντονισμό, διεθνή συντονισμό. Οπότε, για να διδαχθούμε από τα παθήματά μας και να μειώσουμε ε, να αποτρέψουμε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, θα πρέπει να κατανοήσουμε την κατάσταση και να ελέγξουμε τι έγινε με αυτά τα 600 δις ε, δολάρια που κυκλοφορούν στον κόσμο μέσω των παράγωγων προϊόντων. Και αναφέρει και τις ακάλυπτες πωλήσει πριν από λίγο. Θα πρέπει να δούμε, να κατανοήσουμε πώς κυκλοφορούν αυτά τα προϊόντα και να ρυθμίσουμε κάπως την ε, κυκλοφορία τους. Θα πρέπει με αποφασιστικότητα και χωρίς αφέλεια να εγγύψουμε σε αυτό το θέμα. Κύριε Μπούλμαν, σας είπα ότι χρειαζόμαστε τη βιομηχανία για να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία, αλλά θα πρέπει να ε, υποβάλουμε κατάλληλες, σωστές και έξυπνες ρυθμίσεις, ώστε να είναι αποτελεσματικές, γιατί Κάθε λέξη είναι σημαντική. Μόνο έτσι η βιομηχανία μας θα γίνει ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες περιοχές του κόσμου που δεν θα έχουν αντίστοιχα στέρεα θεμέλια. Επίσης έτσι θα καταφέρουμε να προλάβουμε ή να αποτρέψουμε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, αλλά να ρωτήσω το εξή συγκεκριμένα. Θα υπάρξει πρόταση για τα παράγωγα χωρίς εξαιρέσεις, θα υπάρχει οδηγία 4 για τα ίδια κεφάλαια, για τα κυκλικά προϊόντα, τα οποία αξιολόγηθηκαν για παράδειγμα στην Ισπανία και θα δούμε η Ευρώπη να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά ένα χρηματοπιστωτικό φόρο ή άλλα παρόμοια κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίσουν σε θεσμικό επίπεδο ότι οι αιτίε που προκάλεσαν τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα συνεχιστούν. Δεν μπορεί να βοηθάμε τις τράπεζες και στην τελική ανάλυση να μην κάνουμε τίποτα στην χρηματοπιστωτική αγορά, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Η απάντησή μου είναι ναι, κύριε Μπούλμαν. Μετά το ΣΕΡ 3 και χαιρετίζω το ε, έργο της κυρίας Μακάρη, θα έχουμε και την τέταρτη εκδοχή αυτής της οδηγίας στα τέλη του έτους. ΣΕΡ 4 και σίγουρα η οδηγία αυτή θα ασχοληθεί με πολλά θέματα, για τα οποία χρειάζομαι, δώστε μου παρακαλώ λίγες μέρες για να ετοιμαστώ. Μην ε, περιμένετε ε, μεγάλο βαθμό τεχνικής λεπτομέρειας μέσα σε μία μέρα. Χρειάζομαι μήνες για να εξοικειωθώ. Για την ποιότητα ε, των ιδιών κεφαλαίων, για τους κινδύνους ρευστότητας κτλ. Είδαμε τι συνέβη στην Ισπανία με τη, τα δυναμικά αποθεματικά παρόμοια προτάσεις ε, θα εξετάσω και εγώ. Και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί θέλουμε κάποιο βαθμό σύγκλησης στους κανόνες. Thank you very much. Now on behalf of LD... Και τώρα εξ Κύριε υποψήφιε επίτροπε, δεν έχουμε λόγους να αμφισβητήσουμε τη δέσμευσή σας και προσπαθείτε να μας το αποδείξετε, αλλά θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα αρχής, γιατί και εσείς αναφερθήκατε σε αυτή την τάση απομονωτισμού εθνικού που υπάρχει στην Ένωση και ίσως αυτό παρεμποδίσει την βούλησή σας για μεταρρυθμίσεις στην εποπτεία. Και ας μιλήσουμε ε, η, ειλικρινιά ο διορισμό σας οδήγησε σε κάποιε αντιρρήσεις, ιδιαίτερα από την Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιτία τη Εθνικότητά τη. Πολύ αντίθετα έναντι της κοινοτική ένταση. Και η θριαμβολογία του Γάλλου Προέδρου επίσης δεν ήταν πολύ κοινοτικού χαρακτήρα. Και μετά βάλατε ένα γενικό διευθυντή δίπλα σα, ο οποίος επελέγει εξαιτία του διαβατηρία του, ενώ ο προκάτοχός του ήταν ε, εξίσου εισάξιος. Και εξού το ερώτημά μου, γιατί είναι θέμα ουσίας. Επιλέγουμε με βάση το διαβατήριο και την εθνικότητα τα πρόσωπα. Μπορείτε να αντισταθείτε στην ε, γαλλική εξουσία ή των πιέσεων της Βρετανίας. Θα προωθηθεί το κοινοτικό συμφέρον και αυτό γιατί όλος ο κόσμος απαντεί, περιμένει μια ευρωπαϊκή απάντηση και αυτή θα είναι ισχυρή μόνο αν είμαστε ενωμένοι και εργαστούμε για το κοινό συμφέρον. Κυρία Γκουλάρη, πρώτον, ναι, ο κόσμος όλος περιμένει και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να δώσουμε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, και προϊόντων ένα προβάδισμα. Αλλά το ερώτημά σας είναι πολύ σοβαρό, οπότε και εγώ θα απαντήσω πολύ σοβαρά. Τη στιγμή του διορισμού μου άκουσα, διάβασα τα όσα υπόθηκαν. Εδώ και χρόνια πάντω έχω μια κάποια εσωτερική ησυχία, η οποία πλησιάζει το βρετανικό φλέγμα. Πλησιάζει. Δεν τα κατάφερα ακόμα πλήρως σοβαρότερα τώρα. Θα ορκιστώ εάν μου το επιτρέψετε μπροστά στο 10. Και για μένα όταν είναι κανένας Γάλλος πολιτικός άντρα δεν, δεν ορκίζεται συχνά. Αλλά το έχω ήδη κάνει και μπορείτε να ελέγξετε το πώς ε, αυστηρά σεβάστηκα αυτό τον όρκο μου για πέντε χρόνια υποστηρίζοντας το ευρωπαϊκό συμφέρον. Είναι η τιμή μας ως επίτροποι να εκφράσουμε κολεγιακά αυτό το ευρωπαϊκό συμφέρον και να προτείνουμε κείμενα που αυτό επιδιώκουν. Και αυτό είναι ακόμα πιο απαραίτητο όταν βλέπουμε τη βιαιότητα αυτής της παγκόσμιας κρίσης από την οποία πρέπει να εξάγουμε διδάγματα. Μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία κύριε Αγκουλάρ. Ε, είπατε ότι οι προκάτοχοι δεν ήταν ε, λιγότερο εισάξιση. Το αντίθετο, ήταν πάρα πολύ καλή και θα φροντίσω ώστε να αναγνωριστεί το έργο του. Και θα έχω ένα Βρετανό γενικό διευθυντή, αλλά δεν θα είναι Βρετανός, θα είναι Ευρωπαίος. Άλλωστε το έχει αποδείξει και στο παρελθόν και άλλωστε μου έχει ήδη συμβεί να διορίσω όταν πρώτον ήμουν επίτροπο, διόρισα ένα Βρετανό γενικό διευθυντή και ε, καλά περάσαμε και εγώ και αυτό. Δεν είναι ο ίδιο άλλωστε. Όλοι λοιπόν δεσμεύονται από τον ίδιο όρκο να εκφράσουμε το γενικότερο συμφέρον της Ένωσης. Μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα λάβω καμία διαταγή ούτε από το Παρίσι, ούτε από το Λονδίνο, ούτε από οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Έχετε ήδη το χιούμορ αν όχι το φλέγμα. Πιο συγκεκριμένα πάντως για την αποδυνάμωση σε ό,τι αφορά του σχεδίου για την χρηματοπιστωτική εποπτεία που το ΕΚΟΦΗΝ έκανε στην αρχή Δεκεμβρίου. Είχατε μια δήλωση τεσσάρων πολιτικών ομάδων από αυτήν εδώ την ομάδα. Είστε διατεθειμένος να υποστηρίξετε μια κοινοτική λύση και μια ενσωματωμένη λύση που να είναι σωστή για την εσωτερική αγορά ακόμα και αν δυσαρεστήσουν τους μεν και τους δε. Απάντηση. Δεν ξέρω αν έχω χιούμορ, πάντως και σε αυτό το τομέα πρέπει να προοδεύσω. να ένα καλό παράδειγμα αυτού που ονομάζω προστιθέμενη αξία του Κοινοβουλίου που μας χρειάζεται. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο κατέληξε σε μια συμφωνία. Είναι ένα θετικό βήμα. Δεν πρόκειται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε εποπτεία κατά των κυβερνήσεων και των κρατών. Πρέπει μαζί τους να το κάνουμε. Οπότε Περνάω πολύ χρόνο με τους συναδέλφους για να τους πείσω για αυτήν την κοινή φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευαισθησίες. Αλλά στον τομέα αυτό ναι κυρία Γκουλάκ. Δεν θα σας πω εγώ ποιο είναι το αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Ας προσπαθήσουμε να επανέλθουμε προς αυτό το κείμενο. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Thank Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Κόμφεν από τους ε, Πράσινους. Euh. Κύριε Μπαρνιέ, ξανά καλημέρα σας. Πριν την ακρόαση αυτή, άκουσα την ακρόαση του κυρίου Μαγκρίβη, του προκαταχώσου σας. Και υπάρχει κάποιο είδε μια διαφορά στο, στον τόνο. Αυτό που με εκπλήσει πάντως είναι ότι όταν κάνετε τον κατάλογο των οδηγιών που σκοπεύετε να προτείνετε, αναφέρεστε τους τις τέσσερις, αναφέρεται το over the counter, την εποπτεία, μη feed, δηλαδή όλα αυτά τα σχέδια που είναι ήδη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε αυτή η αλλαγή στον τόνο θα συνοδευτεί και από αλλαγή του νομοθετικού έργου και όχι απλώς να επαναλαμβάνετε δεσμεύσεις που είχε ήδη αναλάβει ο προκάτοχος σας. Μιλάμε για φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπου δεν απαντήσατε, Ευρωπαϊκή φορέα για προστασία των επενδυτών όπως της είπα, ε, έλεγχος των φορολογικών παραδείσων. Είναι πολλά από τα θέματα τα οποία δεν θίξατε ακόμα. Απάντηση. Πρέπει να εργαστούμε σοβαρά για θέματα που είναι εξαιρετικά σοβαρά. Για μένα το φίλο μου πορεία είναι πολύ απλό. Είναι αυτό της ομάδας των 20. Και πιο κοντά, μετά από τον προβληματισμό που έκανε ο κύριος Ντελαροζιέρ μετά από αίτημα του Προέδρου Μπαρόζο, για την εφαρμογή και την υποβολή προτάσεων όπως έκανε ο κύριος Ντελαροζιέρ. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για όλη αυτή την νομοθετική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει να κάνουμε παραπάνω, αλλά και καλύτερα. Οπότε ας ξεκινήσουμε και το πρώτο μου τμήμα της θητείας θα είναι να εκπληρώσει σωστά αυτά. μιλήσατε για τη Βασιλεία. Εντάξει, ας τα κάνουμε ήδη αυτά της Βασιλείας, αλλά αυτά είναι ανοιχτά κείμενα και μετά με τις υπηρεσίες μου, εάν γίνω επίτροπος, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε όλα αυτά τα κείμενα. Η η οι, οι φορείς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Και αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο εξετάζουμε. Ε, και η, εργασία του κυρίου Γκοζές, η εποπτεία, αυτό κάνουμε, μη φίδ, αυτό κάνουμε. Ε, ε, θα πάμε ακόμα παραπέρα και με μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα. Ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, παράγωγα προϊόντα, την αντιστάθμιση που είναι βασικός ε, τομέας. Αναφερθήκαμε στις ακάλυπτες πολίτες ε, οψιών τα παράγωγα. Δεν, δεν πρόκειται ε, με τη δικαιολογία του να κάνω μια καλή ακρόαση να σας πω οτιδήποτε. Χρειάζομαι χρόνο. Δεν, δεν είμαι ακόμα διορισμένος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες με τους οποίους πρέπει να έρθω σε επαφή στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι, στη Μαντρίτη, αλλά χρειάζομαι χρόνο πέραν των όσων σας είπα για να οικοδομήσω αυτήν την ατζέντα, αλλά δεν θα αγνοήσουμε κανένα δίδαγμα από αυτήν την κρίση. Κανένα. τι πιστεύετε για το έργο των προκαταγών σας για τις εναλλακτικές πλατφόρμες επενδύσεων στις τράπεζες. Απάντηση, το είδαμε αυτό. Είπατε ότι πολλαπλασιάζονται αυτά στις τράπεζες. Ε, θα το αξιολογήσουμε και μια και θα αναθεωρήσουμε αυτό το κείμενο τους επόμενους μήνες θα σκεφτούμε ένα σωστό τρόπο ελέγχου. Πάντως, το απαραίτητο για να λάβουμε δράση είναι να κατανοήσουμε σωστά. Αυτή τη στιγμή το 85, το 90% αυτών των νέων προϊόντων χρηματοπιστωτικών ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Θα πρέπει όσο γίνεται ευρύτερα να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό. Thank you. Now, on of the ECR. Ευχαριστώ εξ ονόματος του ECR, η κυρία Σφίσμπορν. Ευχαριστώ πολύ, επειδή είμαι η πρώτη συντονίστρια από τη Βρετανία, δεν πρόκειται να ακολουθήσω εθνικές ε, γραμμές. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι πιο πολύ τεχνικό και δεδομένης και της ε, προηγούμενης εμπειρίας σας ως πρώην Επίτροπος και πρώην μέλος του Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργός. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τι θέματα ε, ευθύνης ε, σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα. Ιδιαίτερα Πώς ε, πιστεύετε ότι οι τρεις υποπτικές αρχές, ε, ευρωπαϊκές, θα πρέπει να συνεργαστούν και ποια θα πρέπει να είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που θα πρέπει να είναι μια πλέον αρμόδια. Σε ποιον θα πρέπει να είναι υπόλογη η πρόεδρε του ESA. Και ίσως θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Euh, euh, Απάντηση. Με την κυρία Γκουλάρ προηγουμένως συζητήσαμε το βασικό θέμα της εποπτείας που απορρέει άμεσα από τις συστάσεις του κυρίου Ντελαροζιέρ. Σας είπα ότι είναι τμήμα του φίλου πορεί μας. Αυτές οι αρχές θα έχουν πραγματικές εξουσίες. Θα βασιστούν στις γνώσεις των εθνικών εποπτών εδώ και μερικές εβδομάδες εξετάζω το θέμα και θεωρώ ότι είναι μια σωστή ρεαλιστική λύση να βασιστούμε στους 27 εθνικούς επόπτες σε κάθε τομείς, τραπεζικό, ασφάλειες και αγοράς. Γιατί αυτοί γνωρίζουν τις επιχειρήσεις και τον τομέα τους. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις αρχές που θα σπίζονται. Και σας υπενθυμίζω, όταν δούμε τις Προηγούμενε δομέ που δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο θα είναι οι καινούργιες, το SEPS, ΣΕΙΟΠΣ και CECR, ότι ήδη μεταξύ τους είχαν αυτές οι τρεις ένα μεικτό φορέα που ασχολείται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η Κομισιόν έλαβε στις προτάσεις της υπόψη αυτή την ανάγκη εποπτείας και εδώ έχουμε προβλέψει μια μεικτή επιτροπή που θα πάει παραπέρα των όσων υπάρχουν σήμερα και θα εξασφαλίσει συνεργασία και συνέπεια ανάμεσα στους τομείς αυτό. Τώρα μου λέτε τι θα συμβεί αν υπάρξει μεταξύ τους διαφωνία. Ας δώσουμε ήδη σε αυτούς τους επόπτες δεσμευτικές εξουσίες και αυτό να επιδιώξετε και εσείς να δώσετε σε αυτούς τους επόπτες δεσμευτικές εξουσίες έτσι ώστε σε περίοδο κρίσεως επίγουσα κατάσταση να αναλάβουν δράση, να εφαρμόσουν δίκαια το κοινοτικό δίκαιο να και να ρυθμίσουν τις διαφορές ή διαφωνίες ανάμεσα στους εθνικούς επόπτες. Σε τρία χρόνια θα ξαναδούμε το κείμενο και θα δούμε πώς λειτουργεί, αλλά νομίζω ότι με αυτές τις δεσμευτικές εξουσίες που θα έχουν οι επόπτες θα δούμε πόσο καλά εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ρωτήσω και το εξή. Πολλοί στην Επιτροπή μα έχουν πει ότι θα προτιμούσαν να υπάρχει μια ενιαία υποπτική αρχή στην Ευρώπη. Εσεί θεωρείτε ότι θα ήταν πιο κατάλληλη η μία ενιαία επιτροπή για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα ευθύνη και ποιο είναι υπόλογο σε ποιον. Ε, Αν εννοείται ένα ενιαίο επόπτη που να συγκεντρώνει και τους τρεις επόπτες ανατομέα ή ένας ενιαίος επόπτης που θα καταργούσε τους εθνικούς επόπτες. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι ακριβώς η άποψή σας για το θέμα. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ένας ενιαίος επόπτης. Ξέρετε μια χώρα όπου υπάρχει έτσι. Σε άλλες χώρες υπάρχουν τρεις. Δεν μιλάω για τη ΣΥΠΑ. Δεν υπάρχει πάντως ενιαίο μοντέλο για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι η ποιότητα της εποπτικής δραστηριότητας δεν εξαρτάται απριόρι από την επιλογή. Χρειάζεται εποπτεία και καλή ποιότητα των πληροφοριών εξού και η σημασία της διαφάνειας. Πρέπει να υπάρξει σωστό συντονισμός αυτών των αρχών, σωστή εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών κανονισμών και να ξεκινήσουμε με αυτούς τους τρεις υπόπτες και θα δούμε πώς προχωρούν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Κούβας, ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπαρνιέ, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή ακρόαση. Θέλω να σας πω ότι από τη μέχρι τώρα διαδικασία εκτίμησα την προσπάθεια να δώσετε, να δίνετε σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω τη θέση σας ως μελλοντικού Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών για το θέμα των αποκρατικοποίησεων και ειδικά για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημόσιους οργανισμούς κοινή ωφέλεια για δημόσιες υπηρεσίες. Θα γίνει δηλαδή ανεκτό, όπως έγινε από την πλευρά του προκατόχου σας, του κ. Μαγκρίβη, να γίνονται παρανομίες προκειμένου να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση στην περίπτωση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, όπου για να απολυθεί το πλειοψηφικό πακέτο στην Deutsche Telekom δεν έγινε δημόσια προσφορά εξ όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2004 κάθετος του 25 με συνέπεια να αγνοηθούν τα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων. Σας ρωτώ λοιπόν, θα πάρετε μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας στην προκειμένη περίπτωση. Ε, ε, Κύριε Χουντή, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σεβαστεί τις εξουσίες, την κυριαρχία, την επικουρικότητα στα πλαίσια των κοινών κανόνων μας. Δεν πρόκειται να σας πω ότι θα απαγορεύσουμε, ενθαρρύνουμε ή παρεμποδίσουμε την ιδιωτικοποίηση σε μία ή την άλλη χώρα. Κυβερνήσεις αριστεράς ή δεξιάς είχαν διαφορετικές πολιτικές στα πλαίσια της κυριαρχίας τους από ό,τι βλέπω αναφέρεστε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση στη χώρα σας σε ό,τι αφορά την, την ιδιωτικοποίηση ενός τμήματος των τηλεπικοινωνιών. Άκουσα αυτή την υπόθεση. Ξέρω ότι είχε μεγάλη ηχό στη χώρα σας και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος για τις ανησυχίες σας για την χρηματοδότηση των συντάξεων γιατί όλα αυτά αφορούν το δημόσιο κορβανά και κατανοώ και την ανησυχία για το τι θα μείνει για να χρηματοδοτήσουμε αυτέ τι υπηρεσίε κοινή ωφελία. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη για αυτό το συγκεκριμένη περίπτωση γιατί πρέπει να το μελετήσω περαιτέρω. Αλλά γενικά θα φροντίσω και το είπα αυτό από την αρχή τη ακρόαση και στην ΙΜΚΟ θα έχω συνεχώ τη βούληση να εφαρμόσω σωστό το κοινοτικό δίκαιο και τα επόμενα πέντε χρόνια αν το θέλετε και εσεί. συνεχώς θα προσπαθήσω να προστατεύσω κύριε Χουντή τους μικρούς επενδυτές οι μικροί επενδυτές είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλω να ενισχύσω την πρόσβασή τους στην πληροφορία, στην ενημέρωση και την προστασία. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα θέσουμε επιτάπητος ή θα επαναπροωθήσουμε η τραπεζική κράτα, η, τα δάνεια, το δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό, ακόμα και η εκπαίδευση για οικονομικά θέματα. Αυτό μπορεί να είναι θέμα και άλλων επιτροπών, αλλά κυρίως αφορά και τους πιο ευάλωτους πολίτες. Κύριε Μπαρνιέ και ε, κύριοι συνάδελφοι, αναφέρομαι σε μια περίπτωση που έθιξε τα δικαιώματα 108.000 φυσικών προσώπων, 4.000 νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και ασφαλιστικών ταπείων, Μέρο των εισόδων του είχαν επενδυθεί στον ΟΤΕ. Για αυτά τα δικαιώματα μιλώ. Και επειδή η κοινοτική οδηγία προέβλεπε αυτή τη διαδικασία και δεν ετηρήθη, το πρόβλημα είναι αν εσεί θα πάρετε μέτρα για εφαρμογή αυτή τη κοινοτική οδηγία δεν μιλώ αν θα είναι σωστή ή όχι η αποκρατικοποίηση, τη μορφή αυτή και την κοινοτική οδηγία. Καλό να εφαρμοστεί και εφόσον αυτό είναι σωστό, τότε σα λέω ότι ο σχετικό νόμο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση έχει καταγγελθεί από τη σημερινή ως αντιπολίτευση. Και επομένως έχετε τη βούληση καταρχήν την εθνική να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Euh, Κυρία Χουντή, θα καταλάβετε και θα δεχτείτε την απάντησή μου, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για μια συγκεκριμένη χώρα σε σχέση με μια απόφαση ιδιωτικοποίησης ενός τομέα δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σας δώσω μια απάντηση. Δεν έχω και τα στοιχεία, δεν ξέρω καν αν τα έχουμε και στις μελλοντικέ μας υπηρεσίες αν γίνω ο Επίτροπος. Αλλά η απάντηση είναι ναι, θα φροντίσω στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αυτό θα το κάνω. Θα το συζητήσουμε και με την ελληνική κυβέρνηση και θα φροντίσουμε τη σωστή εφαρμογή. Δεν μπορώ να εκφραστώ διαφορετικά για μια ιδιαίτερη περίπτωση που, αποτά, που απαιτεί εις βάθος ε, απάντηση. Έτσι μπορώ να σας σεβαστώ και ως Ευρωβουλευτή. Αν γίνω επίτροπος θα ε, κοιτάξω τα πράγματα εις βάθος και θα σας δώσω μια απάντηση μετά από μελέτη της περιπτώσεως και για υπό το φως της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Yeah. Σας ευχαριστώ τώρα εξ του ΕΕ, ο κύριος Μπλουμ. Καλησπέρα κύριε Μπαρνιέ. Αναρωτιόμαι μήπως θα μπορούσατε να με καθησυχάσετε λίγο και μιλώ εξ ονόματος ε, της ε, βιομηχανίας του Λονδίνου. Άκουσα τη Δευτέρα το απόγευμα ότι ο κύριος Ρέν δεν ήξερε πως προκλήθηκε η κρίση με τα subprimes και ύστερα άκουσα ε, μία ακρόαση όπου και εσείς τώρα μας λέτε ότι και με ανησυχεί που το, το γεγονό ότι φαίνεται ότι δεν ξέρετε κι εσεί τι γίνεται με τα παράγωγα και με τι ε, πρώτε ύλε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι γίνεται με τις πρώτε ύλε, ότι δεν ε, θα συνεχιστούν τα ίδια προβλήματα. Να θυμόμαστε ότι το 40% του ΑΕΠ ε, της Μεγάλης Βρετανίας προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του Λονδίνου. Να μην ε, σκοτώσουμε λοιπόν τη Χίνα που κάνει τα χρυσά αυγά. Ο κύριος Μπλουμ δεν έφθασε ερώτημα, αλλά εξέφρασε μια πεποίθηση. Έχει το δικαίωμα. Δικός του ήταν ο χρόνος. Και εγώ έχω νούμερα εδώ πέρα για το τι αντιπροσωπεύει το ΣΥΤΙ. Με εντυπωσίαση που είπατε ότι μιλάτε εξ ονόματος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μάλλον μιλάτε εξ ονόματος των, βουλε... των εκλογών σας, των εκλογέων σας. μεταξύ των οποίων υπάρχει μεγάλος αριθμός μισθωτών και στελεχών και εκεί ο κύριος Μπλουμ έχει δίκιο και υπενθυμίζει σωστά ότι για μια μεγάλη πρωτεύουσα όπως το Λονδίνο και για τη Βρετανία είναι σημαντικό το ποσοστό που εκπροσωπούν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είναι σε όλη την Ευρώπη 5 ή 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που σχετίζονται με τον τομέα αυτό. Είναι κόσμος ο οποίος εργάζεται, έχει οικογένειες, αλλά το Λονδίνο είναι η πιο σημαντική αναλογία στη Βρετανική οικονομία είναι η μεγαλύτερη αναλογία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό και θα το προσέξω. Και δεν έχω βεβαίω εδώ την πρόθεση να σας ευχαριστήσω παρά τη θέλησή σας, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι συμφέρον της Βρετανικής χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας, την οποία χρειαζόμαστε όχι μόνο για τη Βρετανία αλλά για όλη την Ευρώπη, δεν είναι συμφέρον της να συνεχίσει να υπομένει όπως εσείς είδατε να γίνει στη Βρετανία γιατί χρησιμοποιήσατε χρήματα του φορολογούμενου και είστε υπόλογος εναντί αυτών για να διορθώσετε τις συνέπειες μιας κρίσης που δεν προεβλέφθη γιατί δεν υπήρχε διαφάνεια, δεν υπήρχε εποπτεία. Αυτή η αγορά των 600 δις που κυκλοφορούν σε όλη τον κόσμο μέσω των παραγόγων προϊόντων πρέπει να ελεγχθεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν κύριε Μπλουμ αυτόν τον έλεγχο. Θα ήθελα εδώ να σας παραθέσω τον Άνταμ Σμιθ απαντώντας που είπε που είναι πατέρας του φιλελευθερισμού. Λέει η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες και χωρίς μια κάποια ηθική αυτό πιστεύω και εγώ. The point I was making Mr. Αυτό που ήθελα να πω κύριε Μπαρνιά και σας ευχαριστώ είναι ότι δεν ζητάω συγγνώμη που εκπροσωπώ το χρηματοπιστωτικό κλάδο του Λονδίνου γιατί χωρίς αυτόν θα ήταν χρεοκοπημένο το Ηνωμένο Βασίλειο και έχω δώσω τις υπηρεσίες μου επί 38 χρόνια. Καταλαβαίνω τι λέει ο Adam Σμιθ και η παράθεση που αναφέρατε, αλλά υπάρχει λάθος νομοθεσία, είναι πάρα πολύ βαριά, είναι πολύ απλά λάθος, είναι πάρα πολύ ακριβή και έχει αποτύχει. Και αυτό που με απασχολεί είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε διδαχτεί τίποτα από το παρελθόν, γιατί φαίνεται να βγάζουμε καινούργια τέτοια νομοθεσία, την ίδια νομοθεσία που απέτυχε στο παρελθόν όπως και στην Αυστραλία για παράδειγμα, δεν ε, υπέστη τέτοιε συνέπειε η Αυστραλία γιατί δεν είχε τέτοια νομοθεσία. Θα κοιτάξουμε λοιπόν άλλα συστήματα νομοθεσία, όχι το σύστημα αυτό το τελείω ε, που, που, θέτει προδιαγραφέ, το οποίο είχαμε ω τώρα και το οποίο προκάλεσε αυτή την επαχτή κρίση. Ε, κύριε Μπλουμ, δεν χρειάζεται να ψάξουμε τα παραδείγματα της Αυστραλίας. Είναι πολύ μακριά την κρίση δεν την εφήβραμε. Είπαμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε, ότι μεταρρυθ... κάνουμε μεταρρύθμιση. Γιατί η κρίση πραγματικά κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική βιομηχανία. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτείτε αυτήν την άποψη που εξέφρασα προηγουμένως. Είναι συμφέρον του της βιομηχανίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να έχει σωστή και αποτελεσματική εποπτεία γιατί έτσι θα έχουμε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες περιοχές του κόσμου. Έχω εδώ ένα άρθρο του Λόρδου Τέρνερ που τον ξέρετε και εσείς και γνωρίζει καλά και τη Σίτη και λέει ότι δεν έμαθε τα διδάγματα της από η, η, η, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρέπει να εξάγουμε διδάγματα από αυτή την κρίση και θα τα εξάγουμε. Από τους μη εγγεγραμμένους ο Χάνς Πίτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε Μπαρνιέ, αποτελείται σημαντικό άτομο και άτομο που έχει ταχθεί υπέρ της Ευρώπης όπως και εγώ, αλλά ασκείται και κριτική σε πολλά θέματα. Χαίρομαι που για σας έχει προβλεφθεί το χαρτοφυλάκιο αυτό τώρα συγκεκριμένα και να εκφράσω την αντίθεσή μου με τον προηγούμενο ομιλητή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να θεωρήσουμε ότι η νομοθεσία, η ρύθμιση προκάλεσε την κρίση αυτή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό παράθεση. Χρειαζόμαστε κανόνες στην οικονομία για κάθε προϊόν, για κάθε τοποθεσία όπου γίνεται εμπόριο και για κάθε θεσμό. Δεν ήμουνα εγώ εδώ έκανε Το θέμα όμως είναι κατά πόσο συμφωνείτε σαφέστατα με αυτή την δήλωση της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ. j'ai Εγώ με δική μου πρωτοβουλία ε, παρέθεσα τα λεγόμενα της καγκελαρίου Μέρκελ για την οποία τρέφω μεγάλο σεβασμό και ήμασταν ταυτόχρονα σχεδόν υπουργοί περιβάλλοντος στις χώρες μας το 94-95 εκείνη στην Γερμανία φυσικά και εγώ στην Γαλλία οπότε άκουσα με ιδιαίτερα προσοχή αυτά που είπε και η κυρία Μέρκελ και ο πρόεδρος Αρκοζή και αυτά που έκανε ο Γκόρντον Μπράουν, ο κύριο Σαπατέρο και άλλοι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στο G20. Βεβαίως, κύριε Μάρτιν, και εγώ είπα ότι καμία χρηματοπιστωτική αγορά, κανένα προϊόν, κανένας φορέας δεν μπορεί να μπει στο απειρόβλητο μιας ε, αποτελεσματικής εποπτείας ε, και μια σωστή επιτήρηση και ελέγχου. Αυτά είπε και στο G20 η κυρία Μέρκελ. Ε, ρύθμιση, ποιοτική ρύθμιση. Αυτό είπα. Και όπως είπε και η κυρία Σαρον χρειάζεται ποιοτική ρύθμιση και αποτελεσματική υποπτία. Και θα πρέπει, χωρίς να κολλησιεργούμε, να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Κύριε Μπούλμαν, πριν από λίγο είπα ότι χρειάζομαι χρόνο για να επεξεργαστώ ένα θέμα που είναι ακαθόδες και πολύ ευαίσθητο και για να υποβάλω προτάσεις, ώστε να προλάβουμε ε, τις επόμενες κρίσεις που αρχίζουν και διαφαίνονται γιατί αρχίζουν και ξαναδημιουργούνται κερδοσκοπικές ποφόλγες. Θέλω να συνεργαστώ με τις τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς για να προβλέψουμε και να προλάβουμε την κρίση. Αν ενσκύψει νέα κρίση, τι σχέδιο εξόδου από αυτήν θα έχουμε. Νομίζω ότι είναι θέμα και φορολογικής ε, φυσικά και δημοσιονομικής κυριαρχίας των κρατών. Αυτό θα το σεβαστούμε. Αλλά προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστώ κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παραστώ και δεν άκουσα τα σχόλιά σας αυτά. Αλλά πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι μεν λένε ότι ε, ήταν πολύ βιαστικό το πακέτο αυτό και ότι δεν είναι εντάξει και οι άλλοι προσπαθούν να το συγκαλύψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και εσείς ε, θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος να εισαχθούν, αν θέλετε, απολομπιστές ε, τροπολογίες, για παράδειγμα, ότι θα προκύψουν ε, επικίνδυνα κενά σε ό,τι αφορά αυτή την πρόθεση που έχετε δηλώσει και που δήλωσε και η κυρία Μέρκελ και τι θα γίνει και από πλευράς Συμβουλίου. Πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε τους συγκεκριμένους σας ε, στόχους και να ασκήσετε συγκεκριμένα πίεση. Κύριε Μάρτιν, μία πρόταση που συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώς θα αντιληθούν συμπεράσματα και διδάγματα από την κρίση. Και υπάρχει το κείμενο, η πρόταση για την εποπτεία, που θα βελτιωθεί. Και το κείμενο για τα hedge funds, ε, για το οποίο έχει έκθεση ο κύριος Γκοζές. Υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες ε, για το θέμα της αποκατάστασης της διαφάνειας και τη ρύθμιση με πολύ συγκεκριμένα και απτά προβλήματα. Τα γνωρίζετε φυσικά. Το θέμα του hedging, αυτό το θέμα της μόχλευσης και ε, το καθεστώς που ισχύει στις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά υπεύθυνοι και αν ε, επικυρώσετε το διορισμό μου, σε συνεργασία με τους συντάκτες ε, και σε συνεργασία μαζί σας, μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Ήδη πρότεινε ο κ. Γκοζές με τα hedge funds και το equity κάποιες προτάσεις. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε αποτελεσματικά και αξιόπιστα κείμενα. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στις ερωτήσεις από τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Θα σας παρακαλούσα να περιορίσετε λίγο το χρόνο μιλία σας. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Λάγκεν. Κύριε Μπαρνιέ, εσείς σε αντίθεση με πολλούς Βρετανούς συναδέλφους είσαστε έμπειρος πολιτικός και ε, πιστός Ευρωπαίος και έχουμε δει ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν κακή η νομοθεσία και ο προκάτοχος Μαγκρίβη επί πέντε χρόνια αρνήθηκε να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Εμείς επιμένουμε όλες αυτές οι υποσχέσεις που έχετε κάνει για καλύτερη και πιο αυστηρή νομοθεσία να εφαρμοστούν. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπατε. Να πω δύο καινούργια στοιχεία. Καταρχάς για τα παράγωγα. Τα παράγωγα είναι 11 φορές μεγαλύτερα από ό,τι το ΑΕΠ πρόκειται για έναν τεράστιο τομέα χωρίς ευθύνη. Έχουμε διδοκοποιήσει ουσιαστικά αυτό το, τα χρήματα που χάθηκαν και έχουμε δημοσιοποιήσει το χρέος. Και το δεύτερο είναι η συμμετοχή του κλάδου, ο συμμετοχή του κλάδου στο κόστος της ρύθμισης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι προτάσεις έχετε να κάνετε, πώς θέλετε να ρυθμίσετε την αγορά των παραγωγών με ευρωπαϊκό τρόπο ή θα περιμένετε μέχρι ότου υπάρξει κάποια ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μια διεθνή νομοθετική ρύθμιση, ακόμη και αν το θέμα αυτό, κύριε Λάγκεν, είναι από τα πιο σοβαρά και σας ευχαριστώ που το θέσατε, γιατί είναι αντίστοιχο με το όγκο των ε, συναλλαγών. Ανέφερα τα 603 εκατομμύρια. Μιλούμε για αστρονομικά ποσά. Μερικές φορές μας φοβίζει και μόνο η σκέψη αυτών των ε, υπέρογκων ποσών. Και στην εντολή του G20 ήδη έχουμε ένα φύλλο Και μια και μιλάμε για το G20, σας είπα και ελπίζω να το καταλάβετε ότι θα αφιερώσω χρόνο και ενέργεια στις συνομιλίε με τους εταίρου μα στην Ουάσιγκτον αρχικά και μετά στην Κίνα γιατί και έχουμε ενδιαφέρουσε εξέλιξεις με την κινέζικη οικονομία. Θα μεταβώ λοιπόν στις χώρες αυτές για να οικοδομήσω σχέσεις και χωρίς να κάνω κηρύγματα και να δίνω μαθήματα θέλω να εξακριβώσω ότι όλοι οι εταίροι μας έχουν αντίστοιχες με εμάς δεσμεύσεις και την ίδια μέρημνα για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και στο Λονδίνο και στο Πίτσμπεργκ. Κύριε Λάγκεν, οι Ηνωμένε Πολιτείε προηγούνται στα θέματα ακάλυπτων πολίσεων, για παράδειγμα. Σε άλλα θέματα, εμείς έχουμε το προβάδισμα. Το θέμα των παραγόγων είναι πολύ σημαντικό. Και επαναλαμβάνω, κανεί να μην βρίσκεται στο πυρόβλητο μια έξυπνη ρύθμιση, όπως ε, λέει η εντολή του G20. Θέλουμε ρύθμιση, εξομάλυνση, τακτοποίηση αυτών των παραγόγων και την θέσπιση κάποιων επιμελητηρίων ε, που θα ασχολούνται με αυτά τα ε, προϊόντα. Υπάρχουν τέτοια συμψηφιστικά γραφεία από αυτά, αλλά ελάχιστα στην Ευρώπη και από αυτά παίρνουν ε, τα παράγωγα προϊόντα. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε τις τάσεις ε, και προς όφελος των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και θα υποβάλω προτάσεις κατά τη διάρκεια του έτους για το θέμα αυτό. Κύριε Μπαρνιέ, δεν έχω διαμορφώσει άποψη για τη συμμετοχή της χρηματοπιστωτικού κλάδου σε ό,τι αφορά το κόστος της του να ξεπεραστεί η κρίση, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι είναι η στάση και είπατε στην αρχή ότι ε, επιμένετε στα ηθικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει και πάλι να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο θέμα αυτό, γιατί χωρίς ε, ευθύνη και σας το λέω απόλυτα πεπισμένος ότι θα πρέπει ο πιστοτικός, χρηματοπιστωτικός κλάδος να προσεγγίσει την πραγματική οικονομία και να μειωθεί και να μην μένουν τα κράτη στο έλεος, αν θέλετε, μιας, ενός κλάδου που έχει χάσει κάθε κατεύθυνση. Θέλετε λοιπόν να εφαρμόσετε αυτούς τις θετικές αρχές. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Φυσικά, φυσικά και ναι. Και μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και αν αποφασίσετε να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θα συναντηθώ με εκπροσώπους ε, των τραπεζών, με εκπροσώπους της ασφάλειας, των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών κτλ. Φυσικά, προετοιμάζουμε το ΣΕΡΔΕ 4 Μίλησε για την ρύθμιση των τραπεζών που θα ενταχθεί στο σύστημα αυτό. Ε, για την ποιότητα των ε, αποθεμάτων, των εγγυήσεων, των ε, ιδίων κεφαλαίων. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να διευκρινιστούν ως απαραίτητες προφυλάξεις για να είμαστε προνοητικοί. Μας ενδιαφέρει αυτό, να είμαστε προνοητικοί. Νομίζω ότι το χρωστάμε στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, στους φορολογούμενους, να κάνουμε μια προσπάθεια έξυπνης ρύθμισης και σε αυτό το θέμα θα εγγύψω ήδη από τις πρώτες εβδομάδες στις θητείες μου, αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Ε, ε, ε, e. Και τώρα η Lulling για το ΕΛΚ. Astrid, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επιτροπέ, θα ήθελα καταρχήν να υποβάλω μια παρατήρηση μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκουλάρη, η συντονίστρια των φιλελευθέρων. Ας μην προβαίνουμε σε δίκη προθέσεων κατά του κυρίου Μπαρνιέ εξαιτία κάποιων θριαβευτικών δηλώσεων που καλό βέβαια ήταν να τις είχε αποφύγει. Καλύτερα λοιπόν να φτάσουμε στο ψαχνό και να σας ρωτήσουμε σε ποιες αρχές θα στηρίξετε τη δράση σας. Φυσικά θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από την κρίση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γιατί με την παγκόσμια αυτή χρηματοπιστωτική κρίση είδαμε να πολλαπλασιάζονται οι διεθνείς φορείς ρύθμισης και η Ευρώπη φαίνεται, όπως και σε άλλους τομείς, θέλει να δώσει, το καλό παράδειγμα. Πολλοί όμως πιστεύουν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τεθεί επικεφαλή σε μια αναδιατύπωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αν όμως διαπιστώσετε ότι οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο πρόθυμοι και δεν διακατέχονται από ένα τέτοιο μεταρρυθμιστικό πάθος, ε, ενώ η ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών στην ε, Ευρώπη υφίσταται τον ε, θέμα ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο θα υπαναχωρήσετε κάπως ε, από αυτή την αφέλεια που δείχνει πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην γίνουμε κορόιδα των άλλων γιατί όπως είπατε 6 εκατομμύρια μισθωτών ε, απασχολούνται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Κύριε Λούλινγκ, δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο αγαθοί στον τομέα αυτό και αφελής. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει φιλοδοξία, να συμπαρασύρει τους άλλους, να αντιλήσει κάποια διδάγματα νωρίτερα τους άλλους, γιατί σε μερικές περιπτώσεις ε, δεν αποθήσαμε από την κρίση. Πάντως έχουμε το προβάδισμα σε θέματα προτάσεων ρύθμισης και εποπτείας και στη θέσπιση κάποιων υπεύθυνων κανόνων για τις αποδοχές των στελεχών, ένα διόλο μελιτέο ζήτημα, ειδικά για τις τράπεζες στις ε, οδηγίες ό,τι αφορά τις απαιτήσει για τα ίδια κεφάλαια. μη φοβάστε με, το, με την πρωτοπορία μας. Δεν νομίζω ότι αυτό θα παραβλάψει την ανταγωνιστικότητά μας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για τον, ε, για ευρωπαϊκό κλάδο και το υπενθύμισε ο κύριος Μπλουμ ο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό Κλάδο έχει την ευκαιρία να βρίσκεται σε μια επικράτεια που θα έχει διδαχθεί από τα παθήματα και θα έχει προβεί σε ρυθμίσεις. Δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια για ένα τέτοιο δεύτερο κλονισμό, τόσου κραδασμούς σαν αυτού που είχαμε στην πρώτη κρίση. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ποιοτικά προϊόντα, γνωστά, ανοιχνεύσιμα. Κυρία Λούλινγκ, το ίδιο ισχύει με τον αγροεπιστημιστικό κλάδο, το ίδιο ισχύει για το κρασί για παράδειγμα και για άλλα προϊόντα. Ε? Μην με παρεξηγείτε, μην με πάρετε με κακομάτι. Χρειαζόμαστε ποιοτικά προϊόντα, να γνωρίζουμε από πού προέρχονται, να είμαστε σίγουροι όταν τα καταναλώνουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Την ίδια ηχνηλασιμότητα θέλουμε και εκεί. Ίσως είναι κάπως τολμηρή αυτή η παρομοίωση, αλλά ξέρετε ότι έχω πάθος με τη ποιότητα της συχνηλασιμότητας. Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Οφείλουμε σεβασμό προς τον καταναλωτή, προς το φορολογούμενο. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε μια παγκόσμια κρίση. Χρειαζόμαστε παγκόσμιες οικουμενικές λύσεις. Και δεν αφιβάλλω ότι οι εταίροι μας που προσυπόγραψαν τις δεσμεύσεις ε, του G20 θα τις στηρίσουν κιόλα. Ευχαριστώ. νομίζω ότι δεν θα έχετε χρόνο για δεύτερη ερώτηση. Χρησιμοποιήσατε το χρόνο σας στην πρώτη ερώτηση. Και να περάσω στον κύριο Κάρας. Κύριε Μπαρνιέ, καλώς ορίσατε και πάλι ως υποψήφιος επιτροπός με πολιτική ηγεσία. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Το Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά της πρόταση του Συμβουλίου για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρόκειται να ακολουθήσει νέα πρόταση για την ενοποιημένη εποπτεία την, όπως ζητάει για το Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερον, στην Επιτροπή της Βασιλείας έχουμε την αίσθηση όλο και πιο πολύ ότι πολλά ευρωπαϊκά κράτη δεσμεύονται και πριν καν υπάρξει νομοθεσία δεσμευόμαστε πώς θα καταφέρουμε το Κοινοβούλιο να κινηθεί παράλληλα και να συμμετάσχει στην Επιτροπή της Βασιλείας και στο G20 πριν από την διαδικασία νομοθεσίας. Πώς μπορούμε να αγγίθουμε τη συνεργασία. Τι προτάσεις έχετε να κάνετε. Euh, Κύριε Καρά, εξ αρχής χαιρέτησα την εργασία που θα πρέπει να κάνετε για την πρόταση για την νέα οδηγία για την απέτηση δύο κεφαλαίων και μιλήσατε για αυτό το νέο πλαίσιο που θα οικοδημήσουμε για την εποπτεία αλλά δεν είμαστε στο τέλος του δρόμου σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Εξέφρασε άποψη το Συμβούλιο και προτιμώ να παρατηρήσω αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη παρά το αντίθετο. Και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου και το Κοινοβούλιο θα δώσει τη δική του προστιθέμενη αξία. Και το είπα και στην κυρία Γκουλάρ, δεν θα πω εγώ οτιδήποτε λιγότερο από αυτό που είπε η φυστάμενη Επιτροπή για την αρχική της πρόταση για τις δεσμευτικές εξουσίες των εποπτών σε αυτούς τους τρεις τομείς έτσι ώστε η γενική αρχιτεκτονική που θα οικοδομήσουμε να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική και θα φροντίσω να συμμετάσχει και το Ευρωκοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Βασιλείας και μια και μιλάτε για την ομάδα των 20 και ο Πρόεδρος Μπαρόζο και άλλοι ηγέτες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, εγώ είμαι διατεθειμένος να σας συναντήσω και εσάς μαζί και με τους άλλους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι και μετά να σας ενημερώσω και στη συνέχεια για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα με αφορούν θα άμασα. Ε, ε, Εκπροσωπείτε αυτή τη Βουλή και στην δική σας Επιτροπή ιδιαίτερα υπάρχει γνώση και πραγματογνωμοσύνη την οποία όλοι αναγνωρίζουν και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και πρέπει να βασιστούμε σε αυτήν για να έχουμε καλούς κανονισμούς. Uh, δεν έχει δεύτερη ερώτηση ο κύριος Καράς και τώρα περνάω στους σοσιαλδημοκράτες και στον κύριο Σκίνερ. Ευχαριστώ, υποψήφια επιτροπέ. Χαίρομαι που καταλαβαίνετε την σημασία ενός ισχυρού χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ευρώπη, είτε στο Φραγκφούρτο είτε στο Λονδίνο, είτε οπουδήποτε αλλού. Γιατί, όπως είπατε και το G20, επισήμανε ότι χρειάζονται αυστηρά ρυθμιστικά πρότυπα για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις που μας πλήττουν. Και κάποιοι επιμένουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι η δύναμη και ελπίζω να το υποστηρίξετε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο σκέλος, αν θέλετε, το διεθνές σκέλος των εργασιών σας, πώς ε, θεωρείτε ότι θα αναπτυχθεί ο ρόλος ε, ισότητας σε ό,τι αφορά θέματα φερεγγιότητας, προκειμένου και οι εταίροι μας να έχουν ίδια επίπεδα νομοθεσίας. Δεν συμφωνείτε ότι θα είναι αποτελεσματική η διεθνής νομοθεσία, γιατί αν δεν υπάρχουν ίσοι όροι θα μειώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και ποιους, ε, ποιες προτεραιότητες θα θέσετε. Κύριε Σκίνερ όλοι εδώ γνωρίζουμε και το λέω για αυτούς που μας ακούν απ' έξω και εδώ ξέρουν γνωρίζουμε το ρόλο που διδραματίζεται ως συντάκτης έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Ασφαλίσεις. Και γνωρίζετε τι συνέπειες μπορεί να έχει εφαρμογή μια σχετική νομοθεσία για τον τομέα των ασφαλίσεων. Όπως είπα και στην προηγούμενη μου απάντηση, έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη κρίση και μια ανίκουστη έξαρση από το 1929. Δεν είχαμε τέτοια κρίση τα τελευταία χρόνια και φυσικά μας ενδιαφέρει και ο διατλαντικός διάλογος κύριε Σκίνερ και με τους μεγάλους μας εταίρους και με την Κίνα γιατί το βάρος της Κίνας και η ισχύ για τους φρύγους της οικονομίας της είναι τεράστια. Θα συνεργαστούμε λοιπόν μαζί της ώστε να συμβαδίσουμε σε πολλά θέματα. Είναι σημαντικός λοιπόν ο παγκόσμιος διάλογος για τα θέματα αυτά. Και για τα λογιστικά πρότυπα είναι πολύ σημαντικό και για τους κανόνες αυτής της προνητικότητας. Γιατί αν θέλουμε καλούς κανόνες και αποτελεσματικούς θα πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να έχουμε ένα κοινό ε, πλαίσιο αναφοράς. Η Deutsche Bank, για παράδειγμα, αν δείτε τον ισολογισμό της με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα ε, ή με τα αμερικανικά, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορές για την ίδια τράπεζα. Ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει, ο ισολογισμός είναι διαφορετικός. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλαίσιο αναφορά ώστε οι κοινοί κανόνε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε όλο τον κόσμο. είπατε ότι χρειάζεται αμοιβαιότητα και για, το, για τη φερεγγιότητα 2. Θα φροντίσω οι αποφάσεις για την αντιστοιχία να στηρίζονται σε μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη αξιολόγηση. Και πιστεύω ότι χάρη στην εργασία μας θα προβούμε σε μια ανεξάρτητη και στιβαρή αξιολόγηση για τα θέματα αυτά. Ένα τελευταίο θέμα για τα λογιστικά πρότυπα και ελπίζω να είναι πλήρης ο ρόλος μας στο Διετραντικό ε, Νομοθετικό Συμβούλιο και θα είναι σημαντικό και εμείς να έχουμε κάποιο ρόλο, αλλά δεν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποιες σωστές αξίες οι οποίες θα προστατεύουν και τους επενδυτές και τους καταναλωτές και όχι μόνο τα, τις τράπεζες και τα βιβλία τους όπως τα βλέπουμε εμείς. Δεν μπορούμε τώρα σε λίγα λεπτά να συζητήσουμε για το θέμα του fair value. Προτιμώ να λέμε market value, αξία της αγοράς παρά δίκαιη αξία, γιατί δεν ταυτίζονται αυτές οι δύο έννοιες. Πάντως για το θέμα των ε, κανόνων θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη μέρημνα της διατήρησης της σταθερότητας και της αποτροπής ε, του κινδύνου μεταβλητότητας που είδαμε πόσο μεγάλη είναι και να κάνω μια σωστή διάγνωση, μια, έχουμε ένα σωστό στιγμιότυπο τη αξία μια επιχείρηση μια δεδομένη στιγμή. Και μαζί στις κύριε Σκίνερ και με άλλους ε, ευρωβουλευτές θα συνεργαστώ για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, φυσικά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό προτιμά η Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να είμαστε και αφελείς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Σας ευχαριστώ και ψάχνω τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Ελκαντράουι. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφιε επίτροπε. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, πολιτική αποζημίωση στην οποία αναφέρατε για τις ε, αποδοχές. Ξέρετε ότι τα συστήματα μπόνους τα οποία συχνά υπολογίζονται στις ε, τα βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα είχαν μοιραία αποτελέσματα. Και φυσικά πέρα από τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο υπάρχει και ένα ηθικό θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το όραμά σας. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις και το 2004 αναφέρεται στις γραπτές σας απαντήσεις ότι θέλετε να προβείτε σε σχετική έκθεση, αλλά φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δεν προχωράμε πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει ευρωπαϊκό, ανάγκη για ευρωπαϊκό πλαίσιο και να υπάρχει κάποια ενιαία διαμόρφωση και αντιολογία στον κλάδο αυτό. Είναι φυσικά αναγκαία η ηθική και η διαντολογία. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Το είπα πριν από λίγο παραθέτοντας και τον Άνταμ Σμιθ. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς το συμφέρον της χρηματοπιστωτικ... του χρηματοπιστωτικού κλάδου κάποιοι κανόνες που θα διέπονται και από ηθική και διοντολογία. Υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάληψης κινδύνου και των υπέρογκων μπόνους και αποδοχών. Πώς τώρα αυτές οι υπερβολικές αποδοχές ενθάρρυναν ορισμένα στελέχη να αναλάβουν ασυλλόγιστους κινδύνους. Νομίζω ότι η δομή των αποδοχών και των πόνους ήταν μία από τις αιτίες της κρίσης. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε διαφανείς κανόνες που δεν θα εθαρρύνουν τέτοια ε, ασυλλόγιστη ανάλυση, ανάληψη κινδύνου ή κοντόφθαλμες ε, και βραχυπρόθεσμες ε, αποφάσεις. Έχουμε και το Financial Stability Board που ασχολείται με τα θέματα αυτά της σταθερότητα και η κυρία Μακάρθη γνωρίζει ότι έχουμε ή πολύ σωστούς κανόνες το ΣΕΡΔΕ 3 που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί για τη διάρθρωση αυτών των αποδοχών και ελπίζω να μπορώ να το πάνω σας για να εγκριθεί από την πρώτη ανάγνωση το κείμενο αυτό. Και κύριε Αρχαντράουι, μακάρι να γίνουμε ακόμη πιο φιλόδοξοι για θέματα της υπευθυνοποίηση των μετόχων. Το ΣΕΡΔΕ που ισχύει για τις τράπεζες και τις ε, επιχειρήσεις επενδύσεων μπορεί να αγγίξει και άλλους τομείς, όπως είναι των ασφαλιών ή των εναλλακτικών ταμείων ε, επένδυσης, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση και τον έλεγχο των αποδοχών. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη δεύτερη ερώτηση. Συμφωνείτε ότι μια τέτοια ρύθμιση, μια τέτοια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για το χρηματοπιστωτικό κλάδο υπό την ευρία έννοια του όρου, αλλά και για όλες τις ε, επιχειρήσεις και όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ειδικά. Νομίζω ότι ήδη απάντησα. Μίλησε για τράπεζες, ασφάλειες, επενδυτικές εταιρείες και εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Άρα η απάντηση είναι καταφατική. it's Mr. Ο κύριος Κλίνς. Κύριε Μπαρνιέ, η βασική, το βασικό, η βασική βλάβη, αν θέλετε, ζημία της κρίσης είναι το πλήγμα στην εμπιστοσύνη στον κλάδο. Και ναι, μεν μπορεί να έχει σβήσει η πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν, ε, υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και υπάρχουν και πρώτες ενδείξεις για προστατευτισμό και επανεθνικοποίηση σήμερα. Και επιπλέον οι καταναλωτές έχουν την εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον κίνδυνο και που προκάλεσαν την κρίση ξεφεύγουν χωρίς να έχουν τιμωρηθεί. Στην ε, Γερμανία απολύθηκε μία υπάλληλος γιατί για ένα μικρό παράπτωμα και θεωρεί ο κόσμος ότι μένουν ατιμόρυτοι υπεύθυνοι της κρίσης. Πώς θα επαναρθώσετε αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αν κάποιοι δεν τήρησαν ε, της ισχύουσης διατάξης υπάρχει δικαιοσύνη που μπορεί να τους ε, διώξει και να τους ε, τιμωρήσει εφόσον υπήρξε παραβίαση νομοθετικών διατάξεων. Τώρα μιλούμε για ένα νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πακέτο που θα αποκαταστήσει την ηθική, τη διοντολογία, θα θεσπίσει κανόνες ε, και θα επαναφέρει κάποιες ευκαιρίε σε αυτό το χρηματοπιστωτικό κλάδο που είναι απαραίτητο για την οικονομία. Η οικονομία χρειάζεται τις αγορές, αλλά θα πρέπει αυτές οι αγορές να υπηρετούν μία υφόρο και ισότιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Είπα κάποια στιγμή στο βήμα στα Ηνωμένα Έθνη, όταν ήμουν υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, αμέσως μετά, μια, μετά στα ηνωμενα εθνη οταν ημουν υπουργο εξωτερικων τη γαλλια αμεσω μετα ομιλία του Μπούς, που είπε να καταστήσουμε ασφαλέστερο τον κόσμο, είπα ασφαλέστερος κόσμος είναι ο δικαιότερος κόσμος. Ο κόσμος σήμερα δεν είναι δίκαιος. Οπότε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει η ανασφάλεια που επικρατεί. Και φέρουμε τεράστια ευθύνη και εγώ ως Επίτροπος, αν μου το επιτρέψετε, και εσείς ως Ευρωβουλευτές, με τις νομοθετικές διατάξεις έχουμε αυτή την ευθύνη να καταστήσουμε δικαιότερο τον κόσμο. Όχι για να υποτιμήσουμε ή να υπονομεύσουμε την οικονομία, αντίθετα για να τις δώσουμε πιο ε, μακροχρόνιες ευκαιρίες, χωρίς ε, δικαιοσύνη, χωρίς ηθική, χωρίς ποιότητα, χωρίς διεντολογία σε αυτόν τον κόσμο, ειδικά για τα τεράστια ποσά ε, ας μην εκπλαγούμε αν ε, ο λαός δεν κατανοεί ή εξεγερθεί. Εγώ θα δώσω μάχη για ένα δικαιότερο κόσμο και θα ήθελα η Ευρώπη να τεθεί στο προβάδισμα αυτού του αγώνα για ένα δικαιότερο κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κλάδος στον οποίο ε, εργαζόμαστε και το χαρτοφυλάκιο σας είναι για τους πιο πολλούς πολίτες ε, κινέζικα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πέρα από το έργο μας, το οποίο θα πρέπει ασφαλώς να κάνουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να δοθεί έτσι ένα κίνητρο για την Ευρώπη. Άλλη μια ερώτηση. Στη Γερμανία υπάρχει ένα ίδρυμα για τον έλεγχο της δοκιμές προϊόντων που κρίνει τα προϊόντα, αν είναι καλά, ικανοποιητικά και το καθεξής. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ισχύσει και για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έχετε κάποια τέτοια ιδέα. Τώρα μιλάτε για την ποιότητα των ειδών διατροφής στην Γερμανία, φαντάζομαι. Όλα τα προϊόντα. Ποιότητα των προϊόντων. Στις χώρες μας όλες. Έχουμε διοικητικές δομές, ε, γραφεία μελετών που εξ ονόματος τους κράτους ε, ελέγχουν την ποιότητα των ειδών διατροφής και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στα σύνορά μας θα πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα των προϊόντων που μπαίνουν στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα προϊόντα που εισέρχονται σέβονται ρήτρε ασφάλειας, αυτά που επιβάλλουμε στους ίδιους τους παραγωγούς μας. Δεν τα λέω με προστατευτικό πνεύμα. Σε ό,τι αφορά πάντως τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, μια και εγώ έκανα ήδη τον παραλογισμό με, για την, απαντώντας στην κυρία Λούλινγκ ανάμεσα στις δύο κατηγορίες προϊόντων, νομίζω ότι πρέπει να εγγυηθούμε στους μικρούς επενδυτές και στους αποτιμιευτές την ασφάλεια των προϊόντων που μπαίνουν στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και μία αρμοδιότητα των εποπτών να ελέγξουν σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Νομίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την ποιότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ο κύριος Γκίγκολτ για τους θα ήθελα να πω το εξή, ότι εδώ στην Επιτροπή μα έχουμε ένα ισχυρό πνεύμα συνεργασία. Γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω δύο ερωτήσει και να λάβω συγκεκριμένε απαντήσει. Πρώτη ερώτηση. Πώ θα διασφαλίσετε ότι ο χρηματοπιστωτικό κλάδο θα πληρώσει το μερίδιο που τον αλογεί για να καλύψει το κόστο στο μέλλον. Δεν έχω λάβει συγκεκριμένη απάντηση και κατά δεύτερον πώς θα διασφαλίσετε ότι στο μέλλον το κοινοβούλιο αυτό θα συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, γιατί στη Βασιλεία, γιατί πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Δεν θέλουμε απλά να επικυρώσουμε, να εγκρίνουμε μια νομοθεσία η οποία θα έχει ληφθεί και θα έχει αποφασιστεί άλλο. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε με βάση και τις αρχές τις οποίες έχετε διατυπώσει και με τις οποίες συμφωνούμε φτάνουμε από ό,τι φαντάζομαι στο τέλος της συνάντησής μας. Και αν θέλετε και εσείς, θα, γιατί από εσάς εξαρτάται, θα είμαι πάντα διαθέσιμος για να συνεργαστώ μαζί σας, να συναντηθώ με εισηγητής, συνεισηγητές και την Επιτροπή σας. Η Κομισιόν σε αυτό το μεγάλο τομέα θα εφαρμόσει το σύνολο των υποχρεώσεων που επιβάλλει η συνθήκη στα πλαίσια της συναπόφασης ε, συνεργασίας ενημέρωσης στις αξιολογήσεις που θα κάνουμε και βεβαίως θα υπάρχει και η τριμερή συμφωνία για την διαθεσμική συμφωνία στην οποία επεξεργάζεται και ο πρόεδρος Μπαρόζο οπότε εγγράφομαι σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος από αυτό και πέρα από την τυπική νομική πτυχή έχω όρεξη να συνεργαστώ μαζί σας να σας ενημερώσω είναι προς δικό μου συμφέρον, δικό σας συμφέρον γιατί γενικά βρισκόμαστε σε συναπόφαση για αυτό για το ερώτημα σας και μετά Είπατε πώς. Δεν τέθηκε το ερώτημα, αλλά μάλλον το, το αναφέρατε. Πώς δηλαδή θα συμμετάσχει ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε μια ιδέα. Η ιδέα ενός φόρου στις συναλλαγές. Η πρώτη ιδέα ήταν του κυρίου Τόμπιν που αναφερόταν σε ένα φόρο στις νομισματικές διακύμανσεις και μετά ε, φόρο στις τράπεζες και γενικότερα στις ε, ροές κεφαλαίων. Αλλά εκεί είναι ένα θέμα. Ποια θα είναι η βάση τη φορολόγησης και μετά σε τι θα χρησιμοποιηθεί είναι το επόμενο ερώτημα. Κάποια κράτη-μέλη θα έλεγαν είναι φόρο για να καταβάλουμε τι δαπάνε που καταβάλαμε να τα βάλουμε στου προπολογισμού και να μειώσουμε το χρέο μα. Υπάρχει πρόβλημα χρέου. Υπάρχει μια άλλη ιδέα την οποία εγώ μπορώ να εκφράσω ως προσωπική άποψη, να δώσουμε το αποτέλεσμα αυτών του, του φόρου για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Με τέτοιου είδους φόρο ίσως να είχαμε πετύχει ένα αποτέλεσμα στην Κοπενχάγη. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Η ανάπτυξη, η, η ένδυα στον κόσμο ή οι, οικολογικέ οικολογικές προκλήσεις. Είμαι, ανοιχτά σε αυτές τις ε, ιδέες. In the στο χαρτοφυλάκιό σας ε, και στις υπηρεσίες σας θα υπάρχουν πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες που θα επηρεάσουν πολύ τα διάφορα νομοθετήματα. Δεν συγκαταλέγονται όμως ούτε ενώσεις καταναλωτών, ούτε συνδικάτα ή τουλάχιστον είναι σε πολύ μικρές ε, μειονότητες και δεν δημοσιεύονται και τα πρακτικά. Θα ήθελα λοιπόν να είναι πιο ίσως και ισορροπημένη η σύνθεση των ομάδων αυτών και να δημοσιεύονται πλήρως τα πρακτικά των συναντήσεών τους. Πρώτα απ' όλα, ο διοικητικό κλάδος που θα διοικήσω είναι υψηλή ποιότητα. Το σύνολο των υπαλλέων συνάντησα πολλούς διευθυντέ, επικεφαλεί των υπηρεσιών και θα είμαι ε, θα είναι τιμή μου να διοικώ τέτοιου είδους ε, διοίκηση. Δεν έχουμε πάντως ε, όλη την γνώση. Γι' αυτό υπάρχουν και επιτροπές, μελέτες και ίσως και ανοίξει αυτές οι, να ανοίξουν αυτές οι, επιτροπές για να είναι καλής ποιότητας πέρα της σωστής ποιοτικής εργασίας που κάνουμε εμείς ως ανεξάρτητη διοίκηση. Και μετά αναφερθήκατε σε επιτροπές που υπάρχουν όπου πιθανότατα υπάρχει μια αναγκαιότητα να ανοίξουν και διαφάνειας. Θα κάνω δηλαδή μια, με επιφύλαξη θετική απάντηση, με την επιφύλαξη του ποια επιτροπή εννοείται. Γιατί δεν μπορώ στην αρχή να σας... Θα ήθελα να συμμετάσχω στη συμφιλίωση της Ευρωπαϊκής ε, της Ενιαίας Αγοράς με τους πολίτες, με τα συνδικάτα, με τις επιχειρήσεις, με τις κοινωνικές δαμές χωρίς να έχουν την εντύπωση ότι εισακούονται πέρα από τη συζήτηση που μπορεί να έχω με την Επιτροπή των Περιφερειών ή της ΕΟΚΕΣ. Δηλαδή είμαι θετικός αυτήν την, το άνοιγμα που προτείνεται. The, uh, Τελευταία ερώτηση από την κυρία Φόρτ από το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπαρνιέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας, ειδικά ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία της οικονομίας. Κανείς δεν θέλει να ζήσει μια κατάσταση όπου θα έχει ξεπολυθεί η παγκόσμια οικονομία και θα έχει έρθει στο χείλος του γκρεμού χάρη σε τέτοιες επικίνδυνες πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πρόεδρος είπε στην αρχή ότι κοιτώντας 50 διαφορετικά νομοθετήματα εδώ στην Επιτροπή αυτή, πολλά εκ των οποίων έχουν να κάνουν για, με την κρίση, για τα μπόνους, τα παράγωγα και το καθεξής. Η ευφυής νομοθεσία θα πρέπει να αποσκοπεί στους, τα σημεία που χρειάζεται και θα πρέπει να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, ακόμα και ο μη θελημένος αντίκτυπος, στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Και το πιο βασικό η πιο βασική κριτική είναι για την AIFM, την ε, σχετική νομοθεσία για τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα οποία θα μπορούσαν να ανέρχονται σε 25 δισεκατομμύρια ανά έτος. Αν καταλαβούμε λοιπόν τον αντίκτυπο αυτό και αν κατανοήσουμε τον αντίκτυπο και των υπόλοιπων 49 νομοθετημάτων, θα εξετάσετε το ενδεχόμενο να τα ξανακοιτάξετε και να τα αναθεωρήσετε τα νομοθετήματα αυτά στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σωστά μαζί. Ε, Ο σκοπός είναι να είναι αποτελεσματικά τα όσα κάνουμε και αν θέλετε κι εσείς θα προχωρήσω σε ένα νέο στάδιο με μεγάλη βούληση γιατί αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Και δεν λέω ότι όλα θα ξεκινήσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπήρξε προηγουμένως πριν την Επιτροπή Μπαρόζο 2 υπάρχουν ήδη μεγάλες νομοθετικές προσπάθειες που θα κληρονομήσω. Ε, σας είπα και ότι από εξ αρχής 1600 νομοθετικά κείμενα διέπουν αυτήν την εσωτερική αγορά. Σε ό,τι αφορά την ευφυή υποπτία των χρηματοπιστωτικών αγορών που επιδιώκω και εγώ βεβαίως και θα έχω την ευκαιρία και με διαφανή τρόπο να αξιολογήσω όλα αυτά τα κείμενα και άλλωστε είμαι διατεθειμένος και το είπα και στην κυρία Μπόλς που έμεινε σε αυτό το έγγραφό της ε, φτάνοντας το είχε δώσει και στον κύριο Αλμούνια. Είμαι διατεθειμένος να το υπογράψω γιατί τίποτα δεν με σοκάρει. Είναι θεμητή η δέσμευση για να κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση για την ε, αξιολόγηση των κειμένων. Για τα hedge funds νομίζω ότι οι κάτοχοι των hedge fund και ο κύριος Γκοζές θα μπορούσε πολύ καλύτερα να τα πει δεν θα πρέπει να φοβούνται αυτού του είδους την νομοθεσία. Είναι προς δικό του συμφέρον. Δεν έχουν συμφέρον να συνεχίσουν να εργάζονται με απουσία διαφάνειας όπως είδαμε στο παρελθόν, να υπάρχουν καλοί κανόνες, να τους σέβονται και ας αναπτύξουν την επιχείρησή τους στα πλαίσια αυτών. Δεν θα αποσύρω πάντως το κείμενο αν αυτό είναι το ερώτημά σας. Στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και να γίνει καλύτερα κατανοητό. Γι' αυτό το κείμενο αυτή είναι η θέση μου για τα hedge fund. Πάντως Συμφωνώ κυρία μου για να κάνουμε μια προσπάθεια για την ποιοτική αξιολόγηση του συνόλου των νομοθετικών κειμένων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δική σας συνδρομή. Thank Σας ευχαριστώ. Η δέσμευση να εξετάσουμε τις ε, μη θελημένες ε, συνέπειες της νομοθεσίας είναι πολύ σημαντική γιατί υποστηρίζουμε τον γενικό στόχο αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες ε, παράπλευρες ε, συνέπειες. Θα μπορούσατε να μας πείτε τις, ε, τα σχετικά πλεονεκτήματα και το πώς θα μπορούσαν αυτό να ευνοήσει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα έχουν και πάλι αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά δεν θα υπόκειται στον έλεγχό μας κάθε ένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αν ο ένας ή ο άλλος βιομηχανικός κλάδος μεταφέρει τις δραστηριότητες του από την Ευρώπη στην άλλη άκρη του κόσμου, γιατί τον υποχρεώνουμε στην διαφάνεια, στην εποπτεία, στο να είναι υπόλογος, αυτοί που θα το κάνουν αυτό, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η δική μου άποψη είναι ότι πέρα από κάποιες παροδικές κινήσεις, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος στο Λονδίνο και αλλού θα κατανοήσει ότι το συμφέρον του θα είναι να βρίσκεται σε μία ήπειρο όπου έχουμε καλούς κανόνες και καλή εποπτεία για να φυλαχθεί αυτός ο οικονομικός κλάδος από όλους τους κινδύνους που είδαμε από τους κραδασμούς και ίσως πιο σοβαρό από την εχθρικότητα των λαών. Θα εξετάσουμε λοιπόν αυτή την ευφυή νομοθεσία. Θα ακούσω τους πάντες. Δεν έχω όρεξη να δημιουργήσουμε την αποδυνάμωση αυτού του οικονομικού κλάδου που χρειαζόμαστε. Αλλά θα μεταρρυθμίσουμε. Θα το κάνουμε με ευφυή τρόπο. Thank you σας ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνονται ο γύρος των ερωτήσεων και τώρα περνάμε στα διαδικαστικά. Θα ήθελα να σας πω ότι οι τρέχουσες αξιολογήσεις για τον ε, υποψηφίων της ΕΚΟΝ θα συνεχιστούν. Η επόμενη συνάντηση είναι στο 5-2 σήμερα στις 8 και αύριο το πρωί στο 1G2 στις 9 το πρωί. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάλκολμ για να ολοκληρώσει τα δικά του διαδικαστικά. Ο κύριος Μπαρνιέ επιθυμεί να κάνει καταληκτικά σχόλια. Έχουμε καθυστερήσει και 10 λεπτά. Μπορώ να σας δώσω όμως ένα λεπτό. Αν θέλετε μπορούμε να μείνουμε εδώ όλο το βράδυ κυρία Πρόεδρε. Θα επανέλθω και αν θέλετε κι εσείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, για την υποδοχή σας προηγουμένως. Κυρία Μπόλς, σημείωσα και την δική σας ανησυχία για μια ποιοτική νομοθεσία. Δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε ως αυτό σκοπό. Το κάνουμε επειδή χρειαζόμαστε καλούς κανόνες για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να προοδεύσουμε. Θα βρίσκομαι πολύ επιτόπου σε αυτόν τον τομέα με τον οποίο εσείς ασχολείστε στην Επιτροπή σας αλλά και στον μεγάλο κλάδο της ενιαίας αγοράς. Σας είπα την πρόθεσή μου μία φορά την εβδομάδα να κάνω τακτικές επισκέψεις σε εθνικές πρωτεύουσες, να συναντώ εθνικές βουλές, συνδικάτα, ενώσεις για να εξηγήσω, για να εξηγώ και να ακούω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σας αν μα θεωρήσετε άξιο και θα ήθελα να προσπαθήσουμε όλοι να ικανοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για την ε, καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ. Uh, Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω και τη συνεδρίασή μας. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή μας ε, έμειναν μέχρι τέλους και αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον μας για τα θέματα αυτά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μπαρνιά για την, τις πολύ συνεκτικές του απαντήσεις και να αναφέρω στα μέλη της Επιτροπής ότι θα τα πούμε στην τεπλανή αίθουσα στις 8. Ευχαριστώ ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του Διερμηνής. Καλό σας βράδυ.